έγκριση τη ημερησία διάταξη είναι το πρώτο θέμα. Σα καλωσορίζω όλου. Διαφωνεί κανεί με το σχέδιο ημερήσιας διάταξη. μήπω έχετε τίποτα σχόλια. Personne. Donc, à défaut... Κανείς. Οπότε θεωρείται εγκεκριμένη ημερήσια διάταξη. Σημείο υπαριθμό 2. Έγκριση των πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων. Δευτέρα και Τρίτη Σεπτεμβρίου και 5 και 6 Οκτωβρίου. Έχετε λάβει και τα πρακτικά ε, ε, αυτά εδώ και λίγο καιρό. Αν έχετε ε, σχόλια, παρατηρήσει, παρακαλείστε να το διαλάσετε στη γραμματεία μέχρι το τη σημερινή συνεδρίαση. Αλλιώ θα θεωρηθούν και τα πρακτικά εγκεκριμένα. ανακοινώσει τη Προέδρου, σημείο 3 δεν υπάρχουν. Ερχόμαστε αμέσως στο σημείο παριθμό 4. Το λόγο θέλει ο κύριος Γιάνσεν, θα το δώσω αμέσως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα μόνο να κάνω μια σύντομη ανακοίνωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την περασμένη εβδομάδα, την 21η Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ε, αρινό λεγόμενο πακέτο, δύο ανακοινώσει. Ένα σχέδιο δράση 12 σημείων πρώτο. Για την υποστήριξη των στόχων της χιλιατίας για την ανάπτυξη και συνοδεύεται αυτή από πέντε έγγραφα εργασίας για την αναπτυξιακή βοήθεια, ε, για εκθέσεις πρόοδο είναι όλες αυτές για το 2010 ε, μία τρίτη για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας. Ένα πρόγραμμα εργασίας 2010-2013 για τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών και ένα πέμπτο έγγραφο αφορά την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης καθώς επίσης και τη φορολόγηση. Όλα αυτά είναι έγγραφα που ονομάζονται staff working paper, έγγραφα εργασία. Έχετε όλα αυτά ε, υπόψη σας και στη διάθεσή σας στην ιστοσελίδα μας. Θα ε, έχει πει και η Επίτροπος άλλωστε. Ευχαριστώ πολύ. Σημείο 5. Δεν έχουμε ε, λάβει ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σημερινή συνεδρίαση, οπότε θα περάσουμε αμέσως στο σημείο υπαριθμών 6. Διαρθρωμένος διάλογος για τις πολιτικές και νομοθετικές προτεραιότητες για το 2011. Ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Κρυσταλία Γεωργίεβα Επίτροπο για τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Αντιμετώπιση Κρίσεων, την οποία και καλωσορίζω. Έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε την κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίευα, Επίτροπο για τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Αντιμετώπιση Κρίσεων. Διαρθρωμένο διάλογο διεξάγουμε για το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011. Ο κύριος Λένε, που είναι πρόεδρος της διάσκεψης των Προέδρων, μας κάλεσε ε, να ε, έχουμε αυτό το διαρθρωμένο διάλογο, ετήσιο διάλογο. Έτσι θα πρέπει να εντοπίσουμε ένα μικρό αριθμό πρωτοφολιών που στη συνέχεια θα διαβάσουμε στον κύριο Λένε. Ε, επισημαίνω ότι πρόκειται για το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011 και όχι για το 2010. Δημοσιεύτηκε αυτό το Μάρτιο, στις 31 Μαρτίου του 2010, στόχος είναι να έχει την ευκαιρία η κυρία Πίτροπος να μοιραστεί μαζί μας ορισμένες σκέψεις για τις προθέσεις της για το 2011 και να μας βοηθήσει να εισφέρουμε και εμείς το προγραμματισμό του 2011 εμ, αναφέροντας ορισμένες από τις προτεραιότητες μας. Έχετε το λόγο κυρία Γεωργίευα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μόνιμη Συγήτρια, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερη χαρά που αισθάνομαι με την ευκαιρία που έχω σήμερα να επανέρχομαι ενώπιόν σας στην Επιτροπή Ανάπτυξης. The work we do, your feedback, your η συμμετοχή δική σας, η καθοδήγησή σας, η ανταπόκρισή σας είναι πάρα πολύ σημαντική για την εργασία μας. Έχουμε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε και όχι οι ευκαταφρόντες. Το πρώτο θέμα σήμερα στην ημερησία διάταξη είναι παρουσίαση των προτεραιοτήτων και του προγράμματο δράσης που ε, εμπίπτουν στη δική μου αρμοδιότητα. Έχουν αλλάξει πολλά από πέρσι που άρχισε να προγραμματίζει για το 2010 την εργασία της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νέο ναι, κοινοβούλιο ανέλαβε, νέα επιτροπή διοριστική και τώρα για πρώτη φορά υπάρχει ξεχωριστός επίτροπος για την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων. Πιο σημαντικό όμως από το θεσμικό πλαίσιο και τις εξελίξεις είναι κάποια άλλα γεγονότα που μεσολάβησαν όπως ε, ε, η τραγωδία στην Αϊτή, η ε, έκρηξη του ηφαιστείου που τόσα προβλήματα προκάλεσε στους εθέρες μας, η πλημμύρη στη Γαλλία με απόλυση ανθρωπίνων ζώων. Και αυτό έφερε πάλι στο προσκήνιο τη δυνατότητα αντιμετώπισης κρίσεων. Γι' αυτούς τους λόγους λοιπόν που σας είπα και τις θεσμικέ αλλαγές αλλά και τα γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο θεώρησα σημαντικό να συζητήσουμε σήμερα για τις προτεραιότητες του 2011 αλλά και του 2010. Ο βασικός στόχος της πολιτικής μου είναι να προωθήσω τη διαδικασία ενίσχυσης της δυνατότητας αντιμετώπισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε στενή συνεργασία με την Κάθη Άστον και άλλους αρμοδίους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δείτε τώρα μια νέα ευκαιρία για να δούμε πώς μπορούμε να συντονίσουμε και να ενισχύσουμε τη δυνατότητα αντιμετώπισης κρίσεων. Ως άμεση συνέχεια στα μηνύματα που μας στέλνει η φύση οι φυσικές καταστροφές, οι θεομηνίες ε, αυξάνονται και ε, στην έντασή τους και στη συχνότητά τους και σε καιρούς ε, δύσκολους δημοσιονομικά χρειάζεται ενισχυμένος συντονισμός και ταχεία απόκριση. Αντίστοιχη ανακοίνωση λοιπόν θα καταθέσω τα τέλη του 2010. Βασικός μας στόχος είναι να αυξήσουμε, να βελτιώσουμε τη ε, δυνατότητα απόκρισής μας σε κρίσεις ε, και αυτή να είναι ταχεία και ορατή. Για να φτάσουμε στο υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας που έχουμε, πάντα με συνένεση, προτίθεμε να Καθοδηγώ αυτή την προσπάθεια, αλλά με συνολική προσέγγιση που θα περιέχει τα εξή στοιχεία. Πρώτον, θα καλύπτει ε, καταστάσεις και εκτός και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν τις κρίσεις στο ιστορικό και πώς στο εξωτερικό της Ένωσης. Δεύτερον, θα αντιμετωπίζουμε τη δυνατότητα ακριβώς ανταπόκρισης κρίσης από ε, διάφορες σκοπιές και με διάφορα σενάρια, όχι μόνο τις πραγματικές καταστροφές και ε, τραγωδίες όπως ε, της ΑΕΤΗΣ που είναι η εξαίρεση μάλλον και παραμένουν και όχι ο κανόνας. Τρίτον, θα εξετάσουμε όλα τα βήματα από την ετοιμότητα Sorry. Συγγνώμη, διορθώνει η Επίτροπος. είμαι λίγο αδιάθετη και παίρνω και φάρμακα. Γι' αυτό καμιά φορά έχω διαλύσεις. Λοιπόν, πρόληψη. Εμ, αντιμετώπιση των κρίσεων, ετοιμότητα. Γνωρίζουμε ότι κάθε σεντ που δαπανούμε για την πρόληψη ε, ε, αυτό στη συνέχεια μεταφράζεται, ε, πολλαπλασιάζεται επί 4 ή μέχρι και επί 10 στην απόδοση που έχει η επένδυση αυτή. Επίσης θα, ε, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμός μεταξύ των τριών πυλών που είναι η πολιτική προστασία, η ανθρωπιστική βοήθεια και η χρήση στρατιωτικών ε, υποδομών όταν αυτό χρειάζεται σε περίπτωση μεγάλων καταστροφών και θεομηνίων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και θέλω ε, όσο γίνεται να είναι ανοιχτό ο διάλογος και να συμμετέχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, να ακούσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια, τα κράτη-μέλη, ανθρωπιστικούς φορείς, προστασία, πολιτική προστασία και οργανισμούς πολιτικής προστασίας βέβαια και τους στρατιωτικούς. Παρένθεση, χθε το βράδυ και σήμερα το πρωί συνεδριάσαμε με τους υπουργούς ε, αμήνης και ήταν πολύ μεγάλη ανταμοιβή αυτό που είδαμε ότι πραγματικά και εκείνοι ενδιαφέρονται, είναι πάρα πολύ προσιλωμένοι στην υπόθεση αυτή και στις αρχές της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ως αποτέλεσμα του διαλόγου αυτού λοιπόν το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει μια νομοθετική πρόταση για την πολιτική προστασία και τα μέσα της, πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις ήδη ε, εφαρμόζονται και μας ε, έχει προτείνει το Κοινοβούλιο τέτοιες δράσεις και τέτοια προγράμματα τα τελευταία χρόνια. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη μου προτεραιότητα. Δεύτερο σημαντικό θέμα για μένα για το 2010 είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και πολλούς από εσάς εδώ παρόντες που συμμετείχαν στην συζήτηση για την ανθρωπιστική ε, βοήθεια. Το 2010 ε, είναι η διάμεση αναθεώρηση αυτής της συνένεσης και του προγράμματος που ε, είναι σε λειτουργία και σήμερα αποτελεί και το σημείο αναφοράς. Επαναλαμβάνω και πάλι σήμερα το πρωί πολλοί υπουργοί εμείς αναφέρθηκαν σε αυτό το μέσο συνεργασίας ως αφετηρία σε περίπτωση αντιμετώπισης κρίσεων αλλά θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε πλέον αυτό το μέσο ως μια ευκαιρία για να προχωρήσουμε. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο, αλλά θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον ή τι ε, διαφορετικό μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Για να είναι ε, όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό. Για να καταθέσουμε και τις σωστές προτάσεις για τις πολιτικές το 2011 και των επομένων ετών. Είναι και η πρώτη ευκαιρία που θα έχουμε να ε, δούμε και τον κανονισμό για να το μελετήσουμε για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ξέρετε ότι ο κανονισμός αυτός ε, είναι το 1996 και εκ τότε δεν έχει τροποποιηθεί ποτέ. Ο κόσμος όμως έχει αλλάξει από το, ε, από το 1996 μέχρι σήμερα και πόσο μάλλον το επόμενο έτη. Θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε και σε ένα σημείο να ενημερώσουμε τον κανονισμό αυτό. Άλλο σημαντικό θέμα και πρωτοβουλία. Νομίζω ότι είναι εδώ κάποιος παρόν που με έχει ρωτήσει και το Φεβρουάριο σχετικά στην ακρόασή μου. Είναι το, το σώμα εθελοντών μάλλον που βασίζεται στο άρθρο 214 της ε, Συνθήκης της Λισαβόνας για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, προγραμματίζουμε για το φθινόπωρο μια τέτοια ανακοίνωση και το θεωρούμε αυτό ένα τρόπο, μια πλατφόρμα ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Όχι μόνο τους νέους εθελοντές, αλλά και νέους επαγγελματίες που ήδη έχουν κάποια εμπειρία και μπορούν να ασχοληθούν με την ανθρωπιστική βοήθεια και να συνεισφέρουν ε, στην επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που τόσο συχνά ε, συμβαίνει στον κόσμο. Υπάρχουν και σήμερα ε, κάποια προγράμματα εθελοντών και προετοιμάζουμε και σχεδιάζουμε στις Βρυξέλλες διάσκεψη για ανταλλαγή απόψεων και βεβαίως θα καλέσουμε και το Κοινοβούλιο να διαδραματίσει ρόλο στη διάσκεψη αυτή. Η ανακοίνωση αυτή που σας έλεγα λοιπόν θα ε, προετοιμάνει το έδαφος για, ε, νόμο, για μια νομοθετική πλαισίωση του 2011 που θα είναι και το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Γνωρίζω ότι υπάρχουν φόβοι στην ανθρωπιστική κοινότητα ε, ότι θα αρχίσουν να κάνουμε τρέλε. Θα παίρνουμε 18χρονου εθελοντέ και θα του στέλνουμε στον κόσμο χωρί να έχουν την επαγγελματική ε, κατάρτιση, εκπαίδευση, την ε, εμπειρία, τη σοφία και την οριμότητα που απαιτείται. Ε, Σα υπόσχομαι ότι θα τηρήσουμε πολύ σοβαρά δύο βασικού κανόνε και αρχέ. Πρώτον, θα έχουμε πρότυπα και προδιαγραφέ επαγγελματικέ που θα πρέπει να τηρούνται για την ανθρωπιστική βοήθεια και δεύτερον, πάντα θα εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και των νέων εθελοντών μας καθώς ε, ε, συστήσουμε το σώμα εθελοντών. Επιτρέψτε μου τώρα να πω σε κάποιες άλλες σημαντικές ε, πρωτοβουλίες για την επιστημιστική βοήθεια και την ανακοίνωση τη σχετική που εκδόθηκε στις 31 Μαρτίου 2010. Γιατί επανέρχομαι, αφού έχει τελειώσει, έχει λήξει, έχει ολοκληρωθεί. Μα γιατί το σημαντικότερο θέμα εδώ στην ανακοίνωση είναι η εφαρμογή της και από ανθρωπιστική σκοπιά δύο πράγματα έχουν πολύ κρίσιμη σημασία. Θα πρέπει να ε, θαρρύνουμε την τοπική ε, επιστηστική βοήθεια. Δηλαδή να μην καταλήξουμε εμείς να τρέφουμε ένα πληθυσμό ε, με εισαγόμενα τρόφιμα καταστρέφοντα την τοπική γεωργία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να είναι ηγετική στην προσπάθεια αυτή, αλλά δεν ακολουθούν και άλλοι. Γι' αυτό θα πρέπει και άλλοι δωρητέ να προσελκυστούν σε αυτή την προσπάθεια και ε, νομίζω ότι είναι πολύ καλός τρόπος, πολύ προοδευτικός και πολύ σόφρον αντιμετώπισης της σιτιστικής βοήθειας. Και θα έρθουμε και στο Κοινοβούλιο ε, να συζητήσουμε την εμπειρία μας στη συνέχεια. Να ζήσετε. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω σε ένα άλλο θέμα συναφές που είναι η πρόκληση για όλους τους δωρητές να συνδέουν την ε, ανθρωπιστική βοήθεια ε, με την ασυγκρότηση. Ε, Στην επιστημιστική βοήθεια, γιατί το λέω αυτό. Όταν δίνουμε επιστημιστική βοήθεια αγοράζοντα τα τρόφιμα επιτόπου, βοηθούμε και την αναπτυξιακή βοήθεια και είναι μια επιπλέον ανακούφιση αυτή. Αυτό είναι μια αρχή που θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας όταν εμείς από την ανθρωπιστική πλευρά ε, έχουμε κάποια δράση ε, επιτόπου για να είναι καλά σχεδιασμένες οι επιχειρήσεις μας. Θα πρέπει να υποβοηθούν και την ανάπτυξη ε, της χώρας αυτής και να συνεργαζόμαστε με τους ομολόγους μας έτσι ώστε να συνδέεται η ανακούφιση της ανθρωπιστικής βοήθειας με ε, την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση των ε, χωρών που υπηρετούμε. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο τελευταίο ε, που είναι η χρηματοδότηση και, ε, και ε, η διαθέσιμη πορεία αλλά και το αν πιάνουν τόπο τα χρήματα που δαπανούμε εκεί. Όπως γνωρίζετε τα από τα δέκα τελευταία χρόνια χρειάστηκε το Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοηθείας ε, έχω να αντλήσει κονδύλια από το αποθεματικό γιατί οι ανάγκες υπερβαίνουν κατά πολύ τη δυνατότητα χρηματοδότησής μας. Και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό και να βγάλουμε και τα αντίστοιχα συμπεράσματα για την κατάλληλη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας ή τουλάχιστον να ε, διευκολύνεται ε, η μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό που έχουμε για τις κατεπίγουσες ανάγκες ε, γιατί σήμερα η διαδικασία είναι πάρα πολύ βαριά και δύσκολη και δεν μπορούμε γρήγορα να αντιδρούμε σε περιπτώσεις και σε χώρες που χρειαζόμαστε επιπλέον οικονομικούς πόρους. Βεβαίως, τούτου λεχθέντος γνωρίζουμε ότι η βασική μα υποχρέωση απέναντι σα και απέναντι στους φορολογούμενους είναι να λογοδοτούμε για το κάθε ευρώ που δαπανούμε, να πιάνει τόπο και να είναι σωστή η δημοσιονομική μας διαχείριση. Τέλος, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τι λησμονημένε κρίσει. Η Επιτροπή σας μας πίεζε πάντα να μην τις ξεχνούμε αυτές. Ε, σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε να ε, προβλέπουμε τουλάχιστον 15% του προϋπολογισμούς μας για τις ε, κρίσεις αυτές, για τις περιοχές αυτές. Ενδεχομένως να έχουμε και νέα κρίση Έχουμε προετοιμάσει κάποιες δράσεις. 24 ε, εκατομμύρια ε, επιπλέον. γιατί γνωρίζουμε ότι ε, επίκυνται και νέε επιστημιστικές κρίσεις και θα χρειαστεί να δοθεί επιστημιστική βοήθεια και σε άλλους. Αυτές λοιπόν οι προτεραιότητές μας. Προσβλέπω στα σχόλιά σα στι υποδείξει σα στι ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Merci Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Οι βουλευτέ έχουν τον λόγο τώρα. Madame Keller. Κυρία Κέλλερ, ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα γιατί μας ενδιαφέρει να ξέρουμε τι επίκειται. Ε, περιλαμβάνει καλές προτάσεις Με ενδιαφέρει να δω ποια στρατηγική θα ακολουθήσουμε για να μην σταματήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά πώς θα τη συνεχίσουμε τόσο ώστε να γίνει πραγματικό εργαλείο για την ανάπτυξη. Δύο ερωτήσεις. Είπατε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εμπλακεί εκ του σύνεγγυ σε αυτή τη διαβούλευση, αλλά και στις υπόλοιπες προσπάθειές σας και στις υπόλοιπες προτάσεις σας. Τι μορφή θα λάβει αυτή η συνεργασία, θα περιμένουμε μέχρι να έρθετε εδώ και να μας προτείνετε ε, να μας παρουσιάσετε δηλαδή τις προτάσεις σας ή αυτή η συνεργασία θα πάρει κάποια άλλη μορφή. Ε, ούτως ώστε να μην μπούμε εμείς, να πείτε εσείς μάλλον εγώ ήρθα και πρότεινα και εμείς πούμε α δεν προτείνατε τίποτα ή θα εμπλέξουμε και τους μη κυβερνητικού οργανισμούς. Δεύτερη ερώτηση. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρξει μια καταστροφή, βλέπουμε ότι έχετε προτάσει για το πώς θα την αντιμετωπίσουμε εσείς και το γραφείο σας, το ιδιαίτερο γραφείο σας, ε, πώς θα δραστηριοποιηθείτε σε άλλους τομείς για την πρόληψη των καταστροφών, ε, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κτλ. Έχετε την αίσθηση ότι θα πρέπει να κάνετε έτσι συγκεκριμένες κινήσεις. Ας απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση. Επίτροπος. Ευχαριστώ. Η πιο σημαντική προτεραιότητα για φέτος είναι η απάντηση στις κρίσεις. Ε, γι' αυτό ακριβώς έχουμε συντάξει ένα έγγραφο και διάφορα σεμινάρια για να το συζητήσουμε. Για να δούμε, για να φτιάξουμε τώρα την ενδιάμεση έκθεση, θα οργανώσουμε και ένα σεμινάριο για να συλλέξουμε απόψεις. Όταν οργανώσαμε τη συζήτηση για την ε, ανακοίνωση, ε, σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε και τα νέα μέσα επικοινωνίας, ε, έναν open forum, ε, δύο, ερωτήσεις, δύο ώρες ας πούμε με ρωταποκρίσεις, ούτως ώστε και αυτοί που είναι απόντες φυσικός πώς να κάνουν τις ερωτήσεις τους. Τώρα, για το σώμα των εθελοντών θα γίνει μια διάσκεψη στις Βρυξέλλες, αλλά θα οργανώσουμε και μικρές ομάδες με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τις εθελοντικές οργανώσεις, για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι μπορούμε να προσφέρουμε, που να έχει σημασία, που να κάνει τη διαφορά. Αν έχετε οποιαδήποτε ε, πρόταση για αυτές τις προτεραιότητες, ε, σας παρακαλώ να δραστηριοποιηθείτε και να πάρετε εσείς την πρωτοβουλία, να έρθετε σε επαφή με το γραφείο μας για να μας έτσι, ενημερώσετε. Εγώ πιστεύω ότι τα σεμινάρια, διασκέψεις ε, που είναι διαρθρωμένες μορφές ε, συζήτησης είναι πολύ καλές για την ετοιμότητα, πρόληψη και την ανταπόκριση. Τον Ιούνιο του 2009 ετοιμάσαμε αυτή τη στρατηγική για τη μείωση των καταστροφών. Αυτή είναι μια καλή βάση που θα μπορούσε να ενσωματωθεί στη νέα στρατηγική για την απόκριση στις κρίσεις. Εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοί μου πιστεύουμε, πιστεύουμε πραγματικά ότι η απάντηση στις κρίσεις είναι, είναι μόνο ένα, από τα τρία σκέλη. Ε, τα άλλα δύο είναι η ετοιμότητα και η συμμετοχή. Αν, ας πούμε, έχουμε μπροστά μας χώρες ε, με ξηρασία, Πρέπει να δούμε τι ανθρωπιστική βοήθεια μπορούμε να δώσουμε, ούτως ώστε οι κοινότητες αυτές οι τοπικές να αφίστανται στην ξηρασία. Αν, ας πούμε, έχουμε να κάνουμε με χώρες, ας πούμε, φτωχέ, που τις έχουν, έχουν πληγεί από τυφώνες. Όταν υπάρχει ανθρωπιστικό πρόβλημα εκεί, καλό είναι να δημιουργήσουμε συστήματα συναγερμού στις χώρες αυτές. Μία τέτοια προσέγγιση προσπαθούμε να προωθήσουμε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και νομίζω ότι μόνο έτσι θα αξιοποιήσουμε και τα λεφτά των φορολογούμενων που δαπανούμε για το σκοπό αυτό. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από τους βουλευτές. Να κάνω εγώ τότε μία ερώτηση. Μιλήσαμε για την οργάνωση αυτού του θελοντικού σώματος, Ευρωπαϊκού Θελοντικού Σώματος για ανθρωπιστική βοήθεια. Τι καθεστώς θα έχει, πώς θα χρηματοδοτείται, πώς θα λειτουργεί αυτό το σώμα ε, και ποιος θα είναι ο ρόλος του δίπλα στις παραδοσιακές ανθρωπιστικές οργανώσεις και φορείς. Κοιτάξτε, είμαστε στην αρχή αυτής της προσπάθειας. προσπαθούμε να δούμε τι δεξιότητες προσόντα θα πρέπει να έχουμε. Είμαστε σε φάση προετοιμασίας για να λειτουργήσει αυτό το σώμα επαγγελματικά. Έχουμε κάνει κάποιες προκαταρτικές επαφές με οργανώσεις εθελοντών και βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και από τα κράτη-μέλη που έχουν δραστηριοποιηθεί και έχουν δημιουργήσει παραδείγματος χάρη τέτοιες οργανώσεις όπως τη Γαλλία. Μίλησα με τον Υπουργό ε, που είναι υπεύθυνο για το Γαλλικό Εθελοντικό Σώμα και ήρθα σε επαφή με διάφορες οργανώσεις που είναι πιο εξειδικευμένες. Παραδείγματος χάρη Medecins Sans Frontières, οι γιατροί χωρίς σύνορα. And, uh, telecom sans Και τηλεπικοινωνίες χωρίς σύνορα, Telecom Sans Frontières. Και μηχανική χωρίς σύνορα. Και τα δύο βασικά μηνύματα που μας στείλανε αυτέ οι οργανώσεις είναι τα εξή. Πρώτον, ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι ξεκάθαρη η εντολή. Το τι θέλουμε να πετύχουμε. Και δεύτερον, να έχουμε και τα λεφτά, ε. Γιατί αλλιώς ξεκινάμε, προσπαθούμε και μετά από δύο-τρία χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Αλλά όπως σας είπα, είμαστε ακόμα στην αρχή. Ελπίζω μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να ξανάρθω εδώ και να σας πω πολύ περισσότερα, πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα για αυτό το σώμα των εθελοντών. Ευχαριστώ η κυρία Κέλλερ ξανά. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να μιλήσω για τις προτεραιότητες, αλλά μια και είσαστε εδώ, ε, ας κάνω μια ερώτηση για την IT. Πόσα από τα, λεπά, από τα λεπτά που υποσχέθηκαν τα κράτη-μέλη ε, στάλησαν όντως στην uh, IT. Ένα δισεκατομμύριο, 234 εκατομμύρια. Είναι εύκολο να μιλήσω για τη δέσμευση της Επιτροπής. Τώρα για τα κράτη-μέλη και για να είμαι δίκαιη, σε πολλά ε, γίνεται συζήτηση αν θα συμμετάσχουν στο Trust Fund των δωρητών ή αν θα δώσουν την υποστήριξή τους στις ε, συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αν θα συμμετάσχουν δηλαδή σε κάποια προγράμματα ή αν θα, συμμετάσχουν σε αυτό το ταμείο, στο trust fund, στο καταπίστευμα. Επομένως δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πού είναι τα χρήματα. Μπορούμε όμως μετά την ε, συζήτηση αυτή να κάνουμε μία επαφή και να σας μιλήσω πιο συγκεκριμένα. Αυτή η ε, συνάντηση που κάναμε για την ε, IT ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ακόμα και πιο φτωχές χώρες ε, προσέφεραν λεφτά για την ΑΕΤ. άρα ξεπέρασε πραγματικά τις προσδοκίες μας αυτή η συνάντηση. Αλλά ανέβασε και τον πύχη. Τώρα έχουμε πραγματικά μπει στο μικροσκόπιο όλου του κόσμου. Ε, για το πού είμαστε. Ε, ο ΙΕ και το Ίδρυμα Κλίντον υποσχέθηκαν ότι θα τους παρακολουθούν όλους όσους δεσμεύτηκαν και θα προσπαθήσουν να βρεθούν τα χρήματα. Και περιμένουν όλοι λοιπόν τα λεφτά που υποσχέθηκε ο Α και ο Β. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω πιο συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορώ να σας μιλήσω για λεφτά. Ο... Η τάδε χώρα τόσα λεφτά. Δεν μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένη. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Πάμε στο σημείο 7. Ας πάμε στην διάσκεψη των δωρητών ε, με τίτλο «Προς ένα καλύτερο μέλλον για την ΑΕΤ» που έγινε στη Νέα Υόρκη στις 31 Μαρτίου του 2010. Εγώ ήμουν επικεφαλής της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας που πήγε ad hoc στο... στη Νέα Υόρκη. Θα σας μιλήσω για τις εντυπώσεις μου. Τώρα όμως θα ήθελα να σας μιλήσω για τις προσωπικότητες που θα συμμετάσχουν σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Καταρχάς θα γίνει η η κυρία Γεωργίευα θα κάνει μια παρέμβαση. Ήταν τμήμα της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μας παρουσιάσει τις δικές της απόψεις και συμπεράσματα. Εν συνεχεία θα ακούσουμε το Ζαζό Ζαν Ιβ, δήμαρχο του Πόρο Θα μας εκφράσει την, άποψη του Δημαρχείου του Πόρο ε, Εν συνεχεία η κυρία Μπενεντίκ Ταρμελά και Μύρτα Κολάρ, Διευθύντρια του Γραφείου ΠΑΜ ε, της ΑΙΤΙΣ. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ε, εξηγήσω λιγάκι ποια ήταν τα απορίσματα της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας Όπω σα έλεγα ήμουν επικεφαλής της αποστολής στη Νέα Υόρκη, ήταν και ο κύριος Γκερέν εκεί. Λόγω του μεγέθου τη της έχει συζητηθεί πολλά το θέμα στο Κοινοβούλιο, κυρίω ε, στην Επιτροπή ε, ε, ανάπτυξη και Ισότιμη σε Χωρών και, και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε αποστείλει διάφορε επιστολέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο Συμβούλιο, ούτως ώστε να ενταχθεί η αποστολή ε, στην, εξωτερική, στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ηγείται η κυρία Άστον, ε, και επίσης ε, του κυρίου Πίμπαλξ και της κυρίας Τζόρτζεβα, που είναι αρμόδια για την ανθρωπιστική βοήθεια και για τη διαχείριση των κρίσεων. για να μεγιστοποιήσουμε την παρουσία της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη, διοργανώσαμε προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις στις 29 και 30 Μαρτίου. Ε, δι συνεδριάσεις, συναντήσεις με την ε, διασπορά από την ΑΕΤ, με τη UNICEF, τη UNDP, τον OCHA ε, και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ε, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία και η Ισπανία συνδιοργάνωσαν αυτή την αποστολή και τελικά για τους 18 επόμενους μήνες έχουμε στη διάθεσή μας 5 5,3 δις. Ε, πολύ περισσότερα από τα 3,9 που ανέμενε η κυβέρνηση της ΑΕΤΗΣ για αυτή την πρώτη φάση της διαδικασίας ε, ανοικοδόμησης. 1,2 δις είναι οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από του πιο σημαντικούς δωρητέ, ε, σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τα 620 εκατομμύρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, και οι συνεισφορέ των κρατών μελών. Η κυρία Άστον τόνισε ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για μια δεκαετία για να ε, παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ και να συμβάλλουμε στην ανοικοδόμηση τη χώρα. Πολλοί ζητούν αλλαγή μεθοδολογία ε, από πλευρά των δωρητών για να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντο. Ε, Κυρίω να υποστηρίξουμε το σχέδιο εθνική αποκατάσταση και ανάπτυξη ε, που είχε προετοιμάσει αρχικά η κυβέρνηση της ΑΕΤ όπου ε, ιεραρχούνται οι διάφορε προτεραιότητες ε, για την ανοικοδόμηση οικονομική, κοινωνική και θεσμική της χώρας και χωροταξική. Επίσης, ε, καλύπτουμε μηχανισμούς ε, συγχρηματοδότηση μέσα στο πρόγραμμα και αναμένεται σημαντική δημοσιονομική βοήθεια και συνεισφορέ ε, από το MDTF, το Ταμείο Πολλαπλών Δωρήτων, που θα διοργανώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κατόπιν θα γίνει η επιλογή των προτεραιοτήτων και θα κατοχυρωθεί μέσα σε ένα πρόγραμμα η συνεργασία και ο συντονισμό των δράσεων όλων των δωρητών. Επίση, προβλέπεται δημιουργία ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα όπου θα αναφέρονται οι αναλήψει υποχρεώσεων από πλευρά των δωρητών. Ε, για να είναι αποτελεσματική συνεργασία, για να κατοχυρωθεί ο συντονισμός. Ε, ε, αναφέρθηκαν πολλές φορές όλα τα επιμέρους σημεία στις συζητήσεις που έγιναν στη Νέα Υόρκη και στα πλαίσια της διάσκεψης αυτής στη Νέα Υόρκη κοινοποιήσαμε τις ανησυχίες που έχουμε ως προς την ανθρωπιστική κατάσταση. Υπάρχουν ακόμη πρόχειροι καταβλισμοί που παρουσιάζουν υγειονομικούς κινδύνους. Πρέπει ταχύτατα να μεταφερθούν από τους καταβλισμούς και πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε καλή ενημέρωση σχετικά ε, με τον τρόπο μεταφοράς αυτών των ανθρώπων για το σχέδιο αποκατάστασης ε, και τις προτινόμενες προτεραιότητες επιμείναμε ούτως ώστε οι τομείς κλειδιά όπως η γεωργία και η επιστημιστική ασφάλεια να μην ε, ε, πέσουν σε δεύτερη μοίρα. Χρειαζόμαστε την ευρύτερη δυνατή διαβούλευση επίσης με την κοινωνία των πολιτών στην ΑΕΤ. Η καταπολέμηση της βίας και της διαφθοράς πρέπει επίσης να αποτελέσουν υψηλή προτεραιότητα για να είναι αξιόπιστες οι δράσεις κυβέρνησης της ΑΕΤΗΣ, Η μελλοντική ε, επιτροπή προσωρινή επιτροπή που θα μετατραπεί στη συνέχεια σε αναπτυξιακό οργανισμό θα αναλάβει βασικό ρόλο για τους δημόσιους διαγωνισμούς, τα δημόσια έργα για να μην υπάρχει και σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς ε, πριν από το σεισμό ούτως ή άλλως υπήρχε μια θεσμική αδυναμία στην ΑΕΤ και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη οικοδομώντας τα νέα προγράμματα. Οπωσδήποτε θα πρέπει τα προγράμματα να συνοδευτούν από μέτρα που θα ενισχύσουν τις θεσμικές δυνατότητες της ΑΕΤ και ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες ε, των τοπικών αρχών ε, γιατί θα εμπλακούν άμεσα στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Η αντιπροσωπεία μας επέμεινε επίσης ούτως ώστε ε, να επικρατήσει διαφάνεια και να γίνει με υπεύθυνο τρόπο η διαχείριση της διαθέσιμης βοήθειας για να έχει η ΑΕΤ τη δημοσιονομική βοήθεια που χρειάζεται αλλά ταυτόχρονα να υπάρξει προσεκτικός έλεγχος ε, κυρίω ω προ τη δημοσιονομική χρήση των κονδυλίων. Επιπροσθέτω, δεν είχαμε πλήρες πληροφορίε για την ίδρυση του Ταμείου που εν μέρη θα διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα, οι όροι λειτουργία αυτού του ταμείου επίσης θα πρέπει να αναλυθούν ενδελεχώς, κυρίως εάν ε, πρόκειται να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτούς τους όρους ε, τη στιγμή που θα ε, δώσει και τη συγκατάθεσή της για τα εν λόγω επιτόπια προγράμματα τακτικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραδείγματο χάρη κάθε τρία χρόνια, να ενημερώνεται για τη διαφανή χρήση των πόρων και για τα πρώτα αποτελέσματα. Η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία θα μεταβεί στην ΑΕΤ τον επόμενο μήνα για να συναντήσει με του φορεί που θα εμπλακούν στη διαδικασία νοικοδόμηση. Ε, και αυτά τα σχετικά έγγραφα ε, ταχύτατα θα μεταφραστούν και στα αγγλικά και θα τα έχετε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ε, τώρα θα αρχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων. Η Επίτροπος έχει το λόγο και στη συνέχεια οι επόμενοι ομιλητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ από την δυναμική αυτής της διαδικασίας, αυτής της διάσκεψης, διακόπτη η Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απλά και ενεργός και στην προετοιμασία και στη διεξαγωγή της διάσκεψης. Η κυρία Στίφλερ συγκεκριμένα ανέλαβε το ρόλο της Προέδρου στη θέση μου κατά τις διμερείς επαφές, ακόμη και στο ε, παρασκήνιο της διάσκεψης. Τώρα, να σας αναφέρουμε ότι στις Βρυξέλλες ε, κάναμε δύο διαβλέψεις με μη κυβερνητικέ οργανώσει που διοργάνωσε ο Επίτροπος Πίμπαλεξε και μία στη Νέα Υόρκη που οργανώσαμε από κοινού με τον ε, κύριο Κλίντον ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει ανέφεραν τα όσα είχαμε συζητήσει στι Βρυξέλλε και τόνισαν το ότι πρέπει να ενισχυθεί η, γεωργική, παραγωγικότητα στο γεωργικό τομέα και ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην επιστημιστική βοήθεια. Πάντως η γενικότερη ιδέα είναι ότι πέρα από την ε, ε, απάντηση που θα δώσουμε, την άμεση απάντηση στην κρίση, πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επέμειναν να έχουμε αυτή την προσέγγιση, δηλαδή πέρα από την ανοικοδόμηση να χρησιμοποιήσουμε την τραγωδία ως ευκαιρία για το μέλλον. Δηλαδή ναι, ε, να ανοικοδομήσουμε τη χώρα, αλλά ε, με βιώσιμο τρόπο. Επίσης, ε, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, ε, ως Ευρωπαία ε, χάρηκα ιδιαιτέρως που εκπροσωπήθηκε σε μεγάλο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν αξιοθαύμαστο. διότι διευκρινίζουμε ποια είναι η θέση μας ε, στην ε, διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια και γενικότερα στη διεθνή σκηνή. Αποδίδω τα εύσημα στα κράτη-μέλη, διότι με τις παρεμβάσεις τους ε, ενίσχυσαν αυτό το αίσθημα αλληλεγγύης που δείχνουμε στην ΑΕΤ και δείχνουμε εμπράκτος πώς θα υποστηρίξουμε την κυβέρνηση της ΑΕΤ, αλλά και προτεραιότητες όπως η αποκέντρωση η ανάπτυξη που στηρίζεται στην δράση των ε, κοινοτήτων, δήμων και κοινοτήτων και οι δράσεις μας ελπίζουμε να ενισχύσουν ε, έτσι περαιτέρω την ΑΕΤ μετά την ανοικοδόμηση θα είναι χρονοβόρα η διαδικασία, αλλά για την ανθρωπιστική βοήθεια και για την αναπτυξιακή βοήθεια θα ήθελα να τονίσω ότι ο χρονικός μας ορίζοντας είναι μία δεκαετία. Αλλά και αυτό κοντόφθαλμο είναι, ξέρετε, γιατί θα χρειαστούμε περισσότερο από δέκα χρόνια. Κοίτα, σας παραπέμπω στην ε, Ανατολική Ευρώπη, στη Βουλγαρία. Συνεχίζεται ε, η μεταβατική περίοδος ε, και αφήστε που ήμασταν πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι όταν κινήσαμε τη διαδικασία σε σχέση με την ΑΕΤ μετά το σεισμό. Οπότε είναι πολύ θετικό που έχουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική και που έχουμε επίγνωση του ότι χρειάζεται βιώσιμη ανάπτυξη ε, και είναι πολύ καλό που προσυπέγραψε αυτή τη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάσκεψη. Δεύτερον, αναλάβαμε άμεσα τη δέσμευση να τηρήσουμε τις ε, ε, υποσχέσεις μας. Ε, θα σας μιλήσω για την Επιτροπή, γιατί μόνο αυτό μπορώ να κάνω. Ο κύριος Επίμπαλξ υπέγραψε πέντε πολύ συγκεκριμένες συμφωνίες. 200 εκατομμύρια για την ανοικοδόμηση της πρωτεύουσας, την ανοικοδόμηση σχολείων, που ε, θα βοηθήσουν πολλά παιδιά. Τρίτον, ε, υποστήριξη της κοινωνίας ε, των πολιτών, όχι με αφηρημένο τρόπο, αλλά με πολύ συγκεκριμένα προγράμματα που έχουν αποδείξει την αξία του σε άλλε χώρε. Τέταρτον, ενίσχυση τη διαδικασία αποκέντρωση ε, σε συνεργασία με ε, το σκέλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολείται με την ανθρωπιστική βοήθεια. Να το εξηγήσω καλύτερα. Εμεί τι κάνουμε. Πηγαίνουμε τη βοήθεια εκεί που βρίσκονται αυτοί που την έχουν ανάγκη. Δεν την συγκεντρώνουμε μόνο στο Πορτοπράζ στην πρωτεύουσα ή σε, σε κάποια άλλη περιοχή. Την πηγαίνουμε εκεί πέρα όπου υπάρχουν ε, πληγέντες γιατί εκείνοι δεν μπορούν να μετακινηθούν. Και ο Επίτροπος επίβαλξε και οι συνάδελφοί μας αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό και ενισχύουν προγράμματα Cash for Job, παραδείγματο χάρη μετρητά εν αντιθέσεων απασχόληση για να αρχίσουν να εργάζονται πάλι αυτοί οι άνθρωποι. Ε, από για την ανοικοδόμηση. Επίσης ε, χρειάζονται και γραφεία για την κυβέρνηση για να ξαρχίσει να εργάζεται αλλά και ανάπτυξη των θεσμικών ε, δογενών ικανοτήτων της ΑΕΤΗΣ. Και από πλευρά των συναδέλφων που ασχολούνται με την ανθρωπιστική βοήθεια σας διαβεβαιώ ότι προσαρμόζουμε τις δραστηριότητες μας σε βάση των άγκων που διαπιστώνουμε επί τόπου. Πάντως ε, θα παραμείνουμε εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστούμε. Ε, ξέρω ότι έχουν την ιδιότητα παρατηρηθεί οι βουλευτές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μα ξέρετε, μας βοήθησαν πάρα πολύ στην αποστολή μας, μας βοήθησαν στη συζήτηση που έγινε για την επισητιστική ασφάλεια. Ε, όπου έπαιξαν ρόλο κλειδί φυσικά και οι μη ε, κυβερνητικές οργανώσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα τον Δήμαρχο του Πόγο Πράνσε Για 10 λεπτά παρακαλώ σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί εμποδίζουν εδώ. Παρακαλώ πάρτε λίγο την κάμερα από <laughs> μπροστά, βλέπουμε τον Δήμαρχο. Ευχαριστώ. Σας έλεγα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε αρμόδια για την ανθρωπιστική βοήθεια, κυρία μόνιμη Συγήτρια για την ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να παρέμβω ενώπιόν σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ε, βασικό θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας ομιλώ στην ειδική συνεδρίαση. Προσωπώ την πρωτεύουσα της ΑΕΤ, Πόρο που είναι σύμβολο τόπος και για την ιστορία, για τον πολιτισμό και για τη ζωή την ίδια των Αιτινών. Έρχομαι ενώπιό σα ως ε, δήμαρχος της 12 Ιανουαρίου του 2010 καταστράφηκε 75% της πόλης αλλά έχω και εντολή από το Δημοτικό Συμβούλιο να σας ε, μιλήσω Ε, και θα πρέπει να σεβαστούμε και να καταλάβουμε την έννοια της ανασυγκρότησης γιατί είναι πολύ της μόδας αλλά πολύ συχνά γίνεται κατάχρηση είναι ε, λαθασμένη αντίληψη που έχει κανείς για την ανασυγκρότηση δεν έχω πολύ χρόνο, μέσα σε 10 λεπτά τι να πω για την ανασυγκρότηση και την ανοικοδόμηση της αίτης ωστόσο θα ήθελα να ε, επισήσω την προσοχή σας σε κάποια βασικά στοιχεία ε, για το ποροπρέν στην πρωτεύουσα και για την ανοικοδόμηση κυρίως θα αρχίσω από τα γενικά και θα περάσω συνέχεια σε ε, πιο συγκεκριμένα. Οικονομικά ζητήματα. Δεν χωράει καμία αμφιβολία και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Η ανασυγκρότηση και νοικοδόμηση της ΑΕΤ, όπως το παρουσιάζει η κυβέρνηση ως θέμα, είναι ε, πρώτα απ' όλα ζήτημα οικονομικό και επενδύσεων και χρειάζονται πολλά χρήματα. Ακούμε υψηλά ποσά στις 31 Μαρτίου οι διεθνείς δωρητές ε, υποσχέθηκαν 9 δισεκατομμύρια δολάρια. 7,2 τα επόμενα χρόνια ήδη είναι κυρίως κρατικές επενδύσεις, ε, δημόσιες, ε, συγχειρίζονται κράτη ή ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, εθνικές ή διεθνείς, ακόμα και, και ιδιωτικές επενδύσεις. όποια όμως και να είναι η εκτέλεση των επενδύσεων αυτών, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ισχύσουν και ορισμένες αρχές που θα καθοδηγήσουν και τη δράση και τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης της ΑΕΤΗΣ. για μας το σημαντικότερο είναι κυριολεκτικά το εξή. Όλες οι επενδύσεις μετά τις 12 Ιανουαρίου του 2010 θα πρέπει να έχουν συμμετοχή έτοιμη κατά 50% τουλάχιστον. Δηλαδή κάθε δολάριο που δαπανάται ως επένδυση ε, στην ανοικοδόμηση της ΑΕΤΗΣ θα πρέπει να έχει συμμετοχή από την IT. Έτσι ορίζει η νομοθεσία μας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση αυτό. Για μας. Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα είναι να ανοικοδομηθούμε από κέντρωση με συμμετοχή και ηγετική ε, δράση της τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι η βασική ε, υπεύθυνοι, οι πρωταγωνιστές, οι εργολήπτες αυτού του έργου. Να φύγουμε από την απλουστευτική αντίληψη που κατηγορεί και ενοχοποιεί τις αρχές και ιδιαίτερα τις τοπικές αρχές. Τώρα είναι μια ευκαιρία να αναζωογονηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση με τους απαραίτητους πόρους και τις απαραίτητες εξουσίες για να εκτελούν τη βασική τους πρώτη αποστολή που είναι η ανακούφιση, και, αλλά η παροχή κοινοφιλών υπηρεσιών επιτόπου και ποιοτικών υπηρεσιών στον πληθυσμό. Παράδειγμα, Πόρο Πράς, ε, η περιφέρεια βούσης. το 12% των ε, κατοικιών που καταστράφηκαν είχαν ε, χτιστεί πριν από το 86. 25% αργότερα και το υπόλοιπο από το 1995 μέχρι το 2000. Η πρωτεύουσα του πόρου ο Πρανς είδε το πληθυσμό της να αυξάνεται από 700.000 το 82 σε 3 εκατομμύρια το 2009. 65% του πληθυσμού ε, ζει σε κατοικίες ε, κακής ποιότητας. 1,5 ε, εκατομμύριο περίπου σε παραγκουπόλεις ζούσαν όπου δεν υπήρχε καμία κοινοφελής υπηρεσία ή πάρα πολύ στοιχειώδες. Τι έγινε μετά τη 12η Ιανουαρίου 2010 στο Πόρο Πράσι. Θα πρέπει να πούμε ότι η πόλη έχει ευκαιρίε. Είναι πάνω στη θάλασσα, ε, έχουν την έδρα του πολλέ κυβερνητικέ υπηρεσίε, πολλέ επιχειρήσει. Είναι σε πλήρη ανάπτυξη ο Δήμος της περιφέρεια τη πρωτευούση ιδιαίτερα. Έχουμε μια πολιτιστική κληρονομιά. 35 ε, γειτονιές με ε, πολίτες που είναι πρόθυμοι να εργαστούν, αλλά ε, έχουν να γίνουν 10 χρόνια εκλογές δημοτικές για τις δημοτικές ε, αρχές. Είναι ευκαιρία τώρα λοιπόν να αναπτυχθεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Μεσολάβησε ε, ο σεισμός και οδηγήθηκε σε παράλυση όλος ο κλάδο τη τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε 300.000 νεκρού, πάρα πολλά θύματα, πολλού ακροτηριασμένου και δυστυχώ πολύ μεγάλε οι ανάγκε και όλε κατεπίγουσε. Πώ αντέδρασε η δημοτική αρχή του Πρέσ. Το Δημοτικό Συμβούλιο επέλεξε να ε, θέσει κάποιους ιδίους στόχους για να βοηθήσει τον πληθυσμό και να διαχειριστεί αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή με ε, συνοδεία και βοήθεια και υποστήριξη στις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις για να μην είναι ε, σκορπισμένη και κατακαιρματισμένη η βοήθεια. Και η ανασυγκρότηση, η ανοικοδόμηση της πόλης. Επίσης θα πρέπει να γίνει αισθητή η παρουσία του κράτους με τη διαχείριση των κρίσεων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, ε, στα, στους καταβλισμούς, στις γειτονιές, με δημοτικούς υπαλλήλους ε, και με ε, κυβερνητικά ε, στελέχη. Γίνεται αυτό τον καιρό μια προσπάθεια καταγραφής και απογραφής του πληθυσμού, παροχή βασικών τροφίμων ως πρώτη και ουσιαστική προτεραιότητα, βεβαίω πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Θέλουμε να καταρτήσουμε μια ομάδα εθελοντών που είναι εξειδικευμένοι ε, στην ανοικοδόμηση. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές μελέτες και πολλές ε, εκθέσεις που κατηγορούν την ανθρωπιστική βοήθεια ότι απαντά μόνο στις επίγουσες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει συντονισμός και τελικά παρεμποδίζεται η μετάβαση ε, σε μια πιο μόνιμη και βιώσιμη ανοικοδόμηση, γιατί είναι αποσπασματική βοήθεια. Η ε, Δημοτική Αρχή επίσης κινητοποίησε την αποκεντρωμένη συνεργασία. Τρέξαμε σε εμπειρογνώμονες για να έχουμε πιο συλλογική δράση, πιο συλλογική αντιμετώπιση. Κοινοτικά κτίρια, δημοτικά κτίρια ως καταφύγια, η ε, πρόθεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των νέων, ιδιαίτερα νέων μηχανικών και σύντομη κατάρτιση ε, στοχευμένη. Ας πούμε, πώς αντιδρά κανείς σε περιπτώσεις ε, θεομηνιών. Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές, ποιες είναι οι σεισμογενείς περιοχές, ποια είναι τα, τα αντισυσμικά υλικά που μπορούμε να χρησιμοποιούμε στις οικοδομές για να περιορίσουμε τη θεομηνία ε, βέβαια ο πληθυσμός πάντα θα παραμένει ευάλωτος. Πολλές από τις μεγάλες πόλεις ε, του κόσμου ολόκληρου ε, αντέδρασαν με αυτή την προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Το Παρίσι, η Μαδρίτη, το Μόντρεαλ και άλλες μεγάλες πόλεις, η Λαροσέλ στη Γαλλία και Διεθνής Ένωση Γαλλοφώνων Δημάρχων πόλεις της Ιβηρικής, ε, Λατινικής Αμερικής και ε, άλλες οργανώσεις ε, δημοτικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε μάθημα σε κανένα, αλλά πρέπει να αποφύγουμε κάποια σφάλματα και να αποφύγουμε και επίγουσα κατακαιρματισμένη δράση. Αυτό δυστυχώς διαπιστώνεται επανειλημμένα, το λένε και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις την τελευταία δεκαετία και σήμερα ακόμα. Πολλές διεθνείς οργανώσεις και ε, ανθρωπιστική δράση στο Πόρο παρεμβαίνουν σε διάφορους τομείς ξεχωριστά. Στην υγεία, στην παιδεία, στην τοπική οικονομία κτλ. Χωρίς ε, ωστόσο να καταλαβαίνουν ότι τα στοιχεία αυτά είναι αλληλένδετα και θα πρέπει να υπάρχει ε, ένα ενιαίο όραμα αντιμετώπισης αυτών των κρίσεων και μια ενιαία θεώρηση. Η ανοικοδόμηση του πόρου πρένσης θα πρέπει να ε, ειδωθεί πάνω από όλους ένα απέραντο εργοτάξιο κυριολεκτικά για την ανάπτυξη την αστική. Ε, συγκεκριμένα θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε στελέχη, επαγγελματίες και εργάτες για όλη τη διαδικασία για να συμμετέχει με τρόπο ενεργό ο πληθυσμός ε, στις δράσεις αυτές για να έχουν συνοχή αποφάσει που λαμβάνονται από τη Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ε, θα ξεκινήσει από ένα στρατηγικό όραμα. με γνώμονα πάντα και τη σύνεση και τη φρόνηση αλλά και μια φιλοδοξία για το μέλλον. Έχουμε μια στρατηγική θεώρηση λοιπόν Έχουμε ε, και πρόταση για τον 21ο αιώνα σε τοπικό επίπεδο, ένα πρόγραμμα δράσης για τον 21ο αιώνα για την ε, βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η ε, Ατζέντα 21 ε, λέγεται ένα άλλο port au prince είναι εφικτό με ε, όσο γίνεται μεγαλύτερη συνεργασία, εταιρική σχέση για να οικοδομήσουμε το μέλλον προς όφελος όλου του πληθυσμού. Βάσει ε, της τοπικής διάγνωσης ε, θα πρέπει να εντοπίσουμε τους στόχους και τα προβλήματα και να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας. Να πρόγραμμα δράσης ή πολλά πρόγραμματα δράσης για να έχουμε κοινό στόχο τη βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη. Όλα αυτά πάντα ε, με αξιολόγηση και έλεγχο των πρόοδων που ε, ε, που έχω. Για το δεύτερο στόχο τώρα, σε μια δεύτερη φάση, από το Μάιο του 2010, θα πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένες δράσεις που να διέπουν όλη την πρακτική με στρατηγικό όρομα, όπως σας είπα, ε, για να ε, υπάρξει περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό εξαρτάται και από τη δυνατότητα χρηματοδότησης για να οικοδομήσουμε μια δημοτική αρχή που να υποστηρίζεται από επιρρογνώμονες μέσα στο επόμενο εξάμεινο. Σημειώστε ότι το Δημαρχείο και τα βασικά ε, δημοτικά κτίρια καταστράφηκαν στις 12 Ιανουαρίου. και άλλε πόλεις είναι στο πλευρό μα και αυτό δείχνει ότι μπορούμε να βγούμε από την κρίση αλλά για να κερδίσουμε αυτή τη σκληρή μάχη για μια βιώσιμη ζωή και μια βιώσιμη πόλη το Δημοτικό Συμβούλιο του Ποροπρένς προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας υποστηρίξει ε, στην ίδρυση ε, του Κέντρου για Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Πρένς. Έχουμε εντοπίσει κάποια στοιχεία που είναι προτεραιότητες στο σχέδιο, η εξήγηση το τι είναι στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, πώς θα επιτευχθεί αυτή με διάδοση της γνώσης και των ε, πρωτοβολιών αυτό παντού σε ε, διασκέψεις και ε, σε όποιον ενδιαφέρεται. Και τέλος, για να για να ανοικοδομήσουμε την ΑΕΤ θα πρέπει να καταλάβουμε τι οδήγησε ε, στην καταστροφή της. Και χρειάζεται να οικοδομηθούν πολλά πράγματα και η ιδιότητα του πολίτη. Πόλη σημαίνει πάνω απ' όλα κοινωνική ζωή, συνύπαρξη, όρεξη για να ζήσει με άλλους ανθρώπους. Η πόλη θα πρέπει να είναι και βιώσιμη και ολοκληρωμένη ως ενότητα. Για μας το πρώτο και βασικότερο είναι η συζήτηση για την οικοδόμηση πρώτα απ' όλα του αιτινού ανθρώπου, του αιτινού πολίτη. Ε, με συνειδητοποίηση, με διαβούλευση. Όπως λέει ο Ροντοβίκ Ζωνά στο κείμενό του για το τσουνάμι που χτύπησε τις 24 Δεκεμβρίου 2004 ε, την Νότια Ανατολική Ασία είναι ε, συνολική προσπάθεια και δημοκρατική. Ε, θα πρέπει να ζητήσουμε επίγουσα ε, αντιμετώπιση των κρίσεων πιο συνειδητοποιημένη και πιο στοχευμένη. Βεβαίως και θα πρέπει να βοηθήσουμε τους πληγέντες και αυτό είναι επίγον αλλά επίσης να είναι για όλους αηφόρα και βιώσιμη ανοικοδόμηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Δημαρχέ. Κυρία Μπενεντίκ πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τις ε, Ευρωπαϊκές Κυβερνητικές Οργανώσεις. Ε, στις 23 ε, Μαρτίου στις Βρυξέλλες δεν ήμουν εδώ, αλλά ήμουν στις 24 Μαρτίου σε μια συνεδρίαση που διοργάνωσαν οι Αμερικανικές ΜΚΟ και στις 25 συν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το γραφείο του Bill Clinton ε, και οι Αμερικανικές μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, οργάνωσαν αυτή την ε, συνεδρίαση. Εγώ εκπροσώπησα τις Ευρωπαϊκές ΜΚΟ και παρουσίασα μαζί με τον Σάμουελ Σίντον που είναι πρόεδρος της Interaction ένα κείμενο κοινό αυτή η, ε, η οργάνωση εκπροσωπεί τις αμερικανικές οργανώσεις. Έχετε αντίτυπα αυτού του κειμένου στην είσοδο. Επικυρώθηκε και από τις αμερικανικές και τις βραζιλιάνικες, χιλιανές, ε, γαλλικές, ε, ισπανικές ΜΚΟ και την Concord. Γιατί οθετήσαμε ένα κοινό κείμενο γιατί οι μη κυβερνητικέ οργανώσει είναι παρούσες στην ΑΕΤ, ήταν και πριν την καταστροφή ε, του σεισμού και κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ, κυρίως αυτέ που ήταν εκεί, αλλά και άλλε οι οποίε ε, δραστηριοποιούνται μετά το σεισμό και αποτελούν μια σημαντική δύναμη για διάφορους λόγους. Καταρχά γιατί παρεμβαίνουν κοντά στον πληθυσμό. Ε, αυτή είναι η προσθέμενη αξία τους. Είναι ότι είναι κοντά στον πολίτη, κοντά στους ανθρώπους. συμμετέχουν ε, σε δραστηριότητες ε, με φορείς ε, της κοινωνίας των πολιτών της ΑΕΤ, τα συνδικάτα των γυναικών, των αγροτών, των οργανώσεων της γειτονιών του Port-au-Prince και επίσης συμμετέχουν και δημόσιες αρχές, δημόσιοι φορείς από την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι τις περιφέρειες, τα διαμερίσματα κτλ. Η ΜΚΟ ε, συγκέντρωσαν 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια για την Ευρώπη. Ε, η συμμετοχή των Ευρωπαϊκών ΜΚΟ ήταν 650 εκατομμύρια. Έχουμε μια έντονη συμμετοχή, γι' αυτό υιοθετήσαμε και αυτή τη δήλωση, η οποία αναφέρει διάφορες αρχές που είναι σημαντικές. Ο Δήμαρχος μίλησε για ανθρωπιστική καταστροφή και μίλησε για την ανάγκη να συντονιστεί το έργο των ΜΚΟ. Ξέρουμε ότι σήμερα σε καταστροφές τέτοιου μεγέθους ε, υπάρχουν πάρα πολλές ΜΚΟ που παρεμβαίνουν και θα πρέπει να συντονιστούμε, να συνεργαστούμε για να αποφύγουμε και τη διασπάθηση αλλά και την, το να κάνουμε τα ίδια πράγματα και να μην ακυρώνουν αυτά που κάνουν κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις κάποιες άλλες. Επίσης, ε, λογοδοτούμε για τις πράξεις μας απέναντι στους ε, με μονομένους ε, δωρητές και χρηματοδότες, βεβαίως τους ε, Ευρωπαίους φορολογούμενους, αλλά και τους ε, δημόσιους δωρητές, τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, απέναντι στις αρχές της ΑΕΤ, λογοδοτούμε και κυρίως απέναντι στον πληθυσμό της ΑΕΤ, γιατί γι' αυτόν δουλεύουμε. Θα πρέπει λοιπόν να συντονίσουμε τις δράσεις μας μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων και με τους ε, χρηματοδότες με τις αρχές της ΑΕΤ και με την κοινωνία των πολιτών της ΑΕΤ. Μία από τις ε, βάσεις ε, της δράσης μας είναι η πρόθεση των δικαιωμάτων, των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών δικαιωμάτων και η πρόθεση των δικαιωμάτων των πιο ευπαθών ανθρώπων, κυρίως των γυναικών, των παιδιών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες ένα από τα βασικά θέματα που τίθενται από το σεισμό και μετά και που θα γίνει όλο και πιο σημαντικό είναι το θέμα της ανοικοδόμησης και την έγκυα δράση. Αν θέλουμε να αναπτύξουμε την γεωργία αν θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα στην ΑΕΤ να εξασφαλίσει την επιστημιστική της ασφάλεια και να κάλυψει τις ανάγκες, θα πρέπει ε, και οι αγρότες και οι γυναίκες και οι πιο φτωχοί, αλλά και αυτοί που μένουν στις διάφορες γειτονίε να έχουν πρόσβαση στις έγκυε προσπάθειε. Όχι όπως να είναι. Ε, υπάρχουν κάποιες ε, περιοχές που δεν θα πρέπει να οικοδομηθούν, αλλά θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει πρόσβαση στη γη. Πρόσβαση στις έγκυες προσπάθειες. Επίσης, θα πρέπει να δυναμώσουμε τους, το δυναμικό των εταίρων μας. Δηλαδή, να προσλαμβάνουμε κυρίως ε, αιτινούς και όχι ξένους, να δώσουμε εκεί προτεραιότητα, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε και πώς τους πληρώνουμε, ούτω ώστε να μην κάνουμε πλειοδοσίες μισθολογικές. Ε, πάντα στις ανθρωπιστικές κρίσεις υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Όταν φτάνουν εκεί ε, μαζικά οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και έχουν τα μέσα και έχουν τα κονδύλια, ε, φτάνουν εκεί διεθνείς οργανώσεις με λεφτά στα χέρια τους, ας πούμε, υπάρχει αυτή η τάση να προσλαμβάνουν άτομα τα οποία θα μπορούσαν να δουλέψουν στην δημόσια διοίκηση της ΑΕΤ. Αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα δημιουργήσουμε δυναμικό ε, στην ΑΕΤ. Θα πρέπει επίσης ε, να κρατήσουμε ένα φυσιολογικό επίπεδο μισθών. Τώρα για να κλείσω αυτό που ακούστηκε στη διάσκεψη της Νέας Υόρκης. Υπάρχει μία εξέλιξη ε, από τις 25 Μαρτίου ε, και μετά. Το γραφείο του ειδικού εκπροσώπου του ΟΗΕ στις 25 Μαρτίου είπε κάποια πράγματα και συνεχεία στις 31 Μαρτίου, μετά τη δήλωση που έκαναν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, βλέπουμε κάποια εξέλιξη στις θέσεις. Ε, έχουμε... Μας καταλαβαίνουν καλύτερα, μας λαμβάνουν υπόψη τους περισσότερο και καταλαβαίνουν τι θέλουμε να κάνουμε. Και εμείς παίρνουμε κάποιες δεσμεύσεις, τις οποίες πρέπει να υλοποιήσουμε. Ε, επομένως, χαίρουμε της εμπιστοσύνης κάποιων ε, αρχών και ελπίζουμε και της ε, κυβέρνησης της ΑΕΤΗΣ. Ε, ζητήσαμε και το κερδίσαμε στην ενδιάμεση επιτροπή για την ανοικοδόμηση της ΑΕΤΗΣ ε, να συμμετέχουμε και εμείς. Πρόκειται για ένα συλλογικό όργανο που θα πάρει αποφάσεις. Εμείς θεωρούσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό ε, ούτως ή άλλως έχει στη διάθεσή του αυτό το όργανο κάποια κονδύλια και θα προωθήσει κάποια αναπτυξιακά προγράμματα. Θέλαμε λοιπόν να είμαστε τμήμα αυτή τη διαδικασία και να συμμετέχουμε σε αυτέ τι αποφάσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Μίρτα Καουλάχ για πέντε λεπτά έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ. Είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. Αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό πράγμα που θέλω να τονίσω είναι ότι πρέπει να αποφύγουμε τον αποκλεισμό. Να υποστηρίξουμε τον ευπαθή πληθυσμό, ε, τους ανθρώπους που δεν έχουν πληγεί, ας πούμε, που δεν έχουν τραυματιστεί από το σεισμό και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτοσχέδιους ε, κατα... καταβλισμού. Αλλά και ανθρώπους οι οποίοι ε, πλήγησαν από το σεισμό και είναι εκτεθειμένοι σε περαιτέρω φυσικές καταστροφές. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πού θα εγκαταστήσουμε τους ε, εσωτερικά εκτοπισμένους μακριά από τις περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή που θα πλημμυρίσουν. Ε, έχουμε ανθρώπους που ζουν τώρα ε, στις όχθες ποταμών που είναι ξερές, αλλά θα έρθουν οι πλημμύρες όπου να είναι. Οπότε προσοχή. Έχουμε άτομα που ζουν στα σχολεία και σε άλλα δημόσια κτίρια που κανονικά χρησιμοποιούνται για την παροχή κοινωνικών και κοινοφιλών υπηρεσιών ή για την για την οικονομική δραστηριότητα. Η προτεραιότητα λοιπόν είναι να επιταχύνουμε την μετακίνηση αν θέλετε αυτών των ανθρώπων, να τους εγκαταστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να έχουμε μια στρατηγική καταφυγίων και να δώσουμε απάντηση στις διάφορες ανάγκες. Ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι άμα τους υποστηρίξουμε μπορούν να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους ε, υπάρχουν όμω και άλλοι άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν καθόλου αυτό, ούτε καν υποστήριξη. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει να δώσουμε βοήθεια για να ε, δώσουμε και βοήθεια εκτό των καταβλισμών, εκεί που ζουν οι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Γιατί ε, πρέπει να προσέξουμε όμως να μην δημιουργήσουμε μια κίνηση ε, ανθρώπων φτωχών που ζουν στις φτωχογειτονιές προς τα, τους καταβλισμούς, ε, δίνοντάς τους την ψευδέστηση ότι εκεί έχουν να κερδίσουν κάτι. Ε, θα πρέπει να δώσουμε βοήθεια εντός και εκτός του Πόγο au επισης Η καταστροφή στο Πόγο au τόσο μεγάλη, τόσο εκτεταμένη, που όλη η προσπάθεια βασικά εστιάζεται στην πόλη. Είναι φυσικό αυτό βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο επίσης να εντοπίσουμε πού ζουν ε, οι εκτοπισμένοι ε, όταν ζουν ε, εκτός του Port-au-Prince. γιατι ζουν σε διάφορες οικογένειες, όχι σε έτσι, αυτοσχέδιους καταβλισμούς. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τοπικά τον κόσμο, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που φιλοξενούν άλλους ανθρώπους εκτοπισμένους, να τους δούμε, να δούμε ποιες είναι αυτές οι οικογένειες, ποιοι είναι αυτοί οι εκτοπισμένοι, να τους βοηθήσουμε, καθώς και τις ευάλωτες κοινότητες που δεν τις έχουμε, που δεν έχουν επηρεαστεί από το σεισμό ούτε από το κίνημα αυτό εξόδου το να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους ε, για να μην επηρεαστούν. Ε, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που επί δεκαετίες δεν έχουν λάβει βοήθεια. Είναι μια ιδιάζουσα πολιτική στιγμή αυτή για την ΑΕΤ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει και εμείς με τη δράση μα να συνεισφέρουμε στον αποκλεισμό. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα τρόφιμα και την ύπαρξη τροφίμων, θα ήθελα να σας μιλήσω για την κατάσταση του λιμανιού του Πχάνσα, που είναι το βασικό λιμάνι εισόδου για τα περισσότερα εμπορεύματα και κυρίως από αυτό το λιμάνι εξαρτάται η χώρα. Το λιμάνι καθώς και ένα μεγάλο τμήμα των αποθηκών του λιμανιού έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό. Μεταξύ του Ιανουαρίου και του Μαρτίου οι εισαγωγές τροφίμων ήταν κάτω από το μέσο όρο και η επισητιστική βοήθεια μάλλον έπαιξε σημαντικό ρόλο για τη σταθεροποίηση των τιμών. Το λιμάνι τώρα είναι το, το πιο ακριβό λιμάνι του κόσμου. Όταν φτάνουν Πιστεύουμε ότι ακόμη και όταν εξομαλυνθεί η κατάσταση, οι τιμέ θα παραμένουν πάνω από τι τιμέ της αγοράς λόγω του προβλήματος με τις υποδομές. Ε, αυτό το κόστο είναι αναπόφευκτο και μπορεί να επιταθεί από κακές καιρικές συνθήκες ε, στην περίοδο των βροχών και τυφώνων. Και αυτό μπορεί να έχει πρόβλημα στην παροχή της τροφής ε, σε όλη την χώρα εμείς ε, ελέγχουμε τις εισαγωγές τροφίμων μαζί με τους εισαγωγείς και αποκινούμε την κυβέρνηση. Προσπαθούμε επίσης να κρατήσουμε ε, ένα αποθεματικό ε, κατεπίγουσας ανάγκης μέσα στη χώρα και η κυβέρνηση σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα με τις εμπορικές ροές θα δει πώς θα το διαθέσει. Τώρα, το Υπουργείο Γεωργίας της ΑΙΤΙΣ προβλέπει ότι η εισοδιά του Ιουλίου, που είναι η πιο σημαντική της χρονιάς, το 2010, θα είναι χαμηλότερη σε σχέση με τη εισοδιά του 2009. Οι σπόροι δεν είναι επαρκείς. Μην ξεχνάτε και τη μετακίνηση του πληθυσμού. Ε, μην ξεχνάτε το γεγονός ότι ο καθένας ε, μοιραζόταν με τους υπολείπους αυτό που έχει, επομένως ε, έχουμε λιγότερους σπόρους. Επομένως, το Υπουργείο ε, Γεωργίας ε, θα κάνουν μια αποστολή τον Ιούνιο για να ε, εξασφαλίσουν, να δουν καταρχάς κατά πόσον υπάρχει, υπάρχουν τρόφιμα σε τοπικό επίπεδο. Θα χρειαστούν χρόνια βέβαια μέχρι να αποκατασταθεί το λιμάνι του Πογοπράς και τα υπόλοιπα λιμάνια και για να, φτάσουν, να φτάσει η γεωργική παραγωγή στα επίπεδα που ήταν πριν από 20 χρόνια. Γιατί μειώθηκε τα τελευταία 20 χρόνια. Ε, πρέπει να γίνει επένδυση για αυτούς τους στόχους. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στο μεταξύ ότι υπάρχει επαρκή στροφή για να υποστηρίξουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο και για να αποφύγουμε την καταστροφή και το χάος. Είμαστε σε μια πάρα πολύ λεπτή κατάσταση τώρα και όταν επενδύουμε σε υποδομές, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει για να υποστηρίξει την πρόσβαση στα τρόφιμα, ε, την επιστηστική ασφάλεια, την ανάλυση, το κοινωνικό δίκτυο, τη γεωργία, την ε, περιβαλλοντική προστασία και τις επενδύσεις στους ανθρώπινους πόρους. Αυτή την ισορροπία θα πρέπει να την διατηρήσουμε. Αν επενδύσουμε σε υποδομές, θα πρέπει παράλληλα να επενδύουμε και στους ανθρώπινους πόρους. Χρειάζεται χρόνος ε, ούτως ώστε ο πληθυσμός ε, να μπορέσει να δρέψει τους καρπούς από αυτές τις επενδύσεις ε, που κάνουμε. Ο κόσμος χρειάζεται τώρα κάτι. Και αυτό μπορούμε να, το, να πετύχουμε, μπορούμε να πετύχουμε να εξασφαλίσουμε αυτήν την ισορροπία εάν επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αρχίσουμε τις ερωταπαντήσεις τώρα. Ο κύριος Μίτσελ θα πάει πρώτος στο λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που μας αφιέρωσαν το χρόνο του σήμερα. Ευχαριστώ όλους ιδιαίτερα στο Δήμαρχο του Πόρτο Πράνσε. Ούτε να φανταστούμε δεν μπορούμε το πόνο αυτών των ανθρώπων ε, και σας ευχαριστούμε για την έκθεσή σας, ε, Πρόεδρο, και που υγείστε τις αντιπροσωπείες. Ε, την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή συζήτησα εν συντομία το θέμα με την Επίτροπο για αυτό το εγχειρίδιο για την ανοικοδόμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο πρέσβης της ΑΕΤ ε, ε, ήταν στην ίδια συνεδρίαση με μένα πριν από δύο μήνες, αν θυμάμαι καλά, όταν συζητήθηκε αυτό το εγχειρίδιο. Μα να μην επανεφεύρουμε τον τροχό, έτσι, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε στην διαδικασία νοικοδόμησης θα χρησιμοποιήσουμε αυτά που ήδη έχουμε. Θα συνεργαστεί η Επιτροπή με την ε, κυβέρνηση της ΑΕΤΙΣ και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, της ΑΕΤΙΣ για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εγχειρίδιο που ήδη υπάρχει. Δεν, πρόλαβε, δεν ε, προσγειώθηκε το αεροπλάνο μου εγκαίρος και δεν τα άκουσα όλα, ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Αυτό που θέλω να μάθω είναι το εξής. Ε, στο Πόρτο Πράνση γενικότερα στην Αιτία έχω την εντύπωση ότι έχει εκτοπιστεί μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και από ό,τι κατάλαβα μπορούν ναι, να επιστρέψουν κάποιοι, αλλά μήπως απομονωθούν να επιστρέψουν ε, ε, στις, στα χωριά τους. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να εγγυηθούμε την ασφαλή επιστροφή αυτών των εκτοπιστέντων. Επίσης, μία ερώτηση προς τον Δήμαρχο του Πόρτο Πράνς. Ε, ενίοτε ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ είναι ε, η ιδιοκτησία. Χρησιμοποιούμε εμείς, παραδείγματος χάρη, τις δορυφορικές εικόνες μας μετά το τσουνάμι, Φερρυπίν, ε, στη Ταϊλάνδη και σε άλλες περιοχές του κόσμου για να βοηθήσουμε κάποιους για τον εντοπισμό των ιδιοκτησιών τους ε, ε, για να εντοπίσουν κάποια αγροτεμάχια. Είτε πρόκειται να τα αφήσουν μετά για γρανάβευση, να τα χρησιμοποιήσουν. Τι γίνεται λοιπόν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς για έγκαιη ιδιοκτησία μιλώ, στην ΑΕΤ. Είναι δυσχερέστατες οι συνθήκες, ε, πολλοί δεν είχαν αγροτεμάχια. Μήπως τώρα μπορούμε να προάγουμε την έγκαιη ιδιοκτησία. Μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό. Όχι να έχουμε μόνο τους σπόρους και την καλλιέργεια. Να χρησιμοποιηθεί αυτό το κεφάλαιο. Ε, στο 19ο αιώνα στη δικιά μου τη χώρα αυτό κάναμε και ε, ε, γιατί στην Ιρλανδία έγινε κατανομή της γης και χρησιμοποιήθηκε ως ε, κεφάλαιο η η ιδιοκτησία και δεν καλλιεργήθηκε απλώς με επιμορτία. Δεν θεωρείτε ότι είναι καλή ιδέα να ενισχύσει αυτή την προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, ε, θα πρέπει να έχουμε μια ε, συνολική προσέγγιση, δηλαδή ολόκληρη η νήσος. Τι έγινε στη Δομινικανή Δημοκρατία, ποιες απώλειες υπήρχαν εκεί. Μήπως Θα μπορούσαμε να είχαμε μια ε, καλύτερη κατανομή των απολειών αν υπάρχει καλύτερη συνεργασία σε ολόκληρο το νησί. Ε, και τελευταία ερώτηση. Ε, πώς θα γίνει, Πρόεδρε, να, παραμείνουν, να παραμείνει το φως της δημοσιότητας σε αυτό το πρόβλημα, γιατί πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα υπάρχουν. Πώς θα ανταποκριθούμε με βιώσιμο τρόπο. Ε, ευχαριστώ και σταματώ εδώ για να έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Υπάρχουν ε, άλλε ερωτήσεις. Ε, θα ήθελε κάποιο άλλο το λόγο. Ο κύριο Μαρτίνες. Ευχαριστώ πολύ. Διάβασα βεβαίω με πολύ, άκουσα συγγνώμη με πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπατε και εσεί οι ίδια στη συνέχεια την κυρία Επίτροπο και ιδιαίτερα τον εμπειρο, τους εμπειρογνώμονές μας. και το δήμαρχο του Ποροπράς. Και είναι πάρα πολύ τιμα αυτά που μας είπε. Και πολύ σωστά. Πολύ σωστός ο, προ... προσανατολισμός που σκιαγραφεί ο Δήμαρχος μέσω της παρουσίασής του. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι Όλο όσα φανταζόμαστε για την οικοδόμηση της ΑΕΤΗΣ, όπως θα τα φανταζόμασταν για την ανοικοδόμηση της οποιασδήποτε χώρας που είχε καταστρο... καταστραφεί μετά από ένα τέτοιο πλήγμα. Όλα αυτά εξαρτώνται βεβαίως από τις ίδιες τις δομές της χώρας. Το πρόβλημα που θεωρώ ότι υπάρχει στην ΑΕΤ, όσο γνωρίζω την, την ΑΕΤ, είναι ότι είναι μια χώρα που δεν έχει πραγματικές και σταθερές ε, δομές. Το λέω πραγματικά ομά και καθόλου διπλωματικά. Όπως είχαμε πει σε μια προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, υπήρξαμε μάρτυρας δύο μεγάλων σεισμών. Σε ένα διάστημα εβδομάδων θα έλεγα. Σε μια χώρα στην Αϊτή καταρχήν, όπως η Αϊτή, και εν συνεχεία σε μια χώρα όπως η Χιλή. Η μεγαλύτερη διαφορά στις δύο περιπτώσεις είναι ότι έχουμε ένα κράτος από τη μία που έχει δομές, ένα κράτος που έχει δομές σταθερές και έχουμε και από την άλλη μια άλλη χώρα όπου οι κρατικές δομές και η κοινωνία είναι σχεδόν ξεχαρβαλωμένες. Και νομίζω ότι αυτό που συζητάμε τώρα, αυτό που μαντεύω από τα λόγια του Δημάρχου είναι ότι πρέπει να κάνουμε την ανοικοδόμηση όχι για να ανοικοδομήσουμε αυτό που δεν υπήρχε, αλλά να οικοδομήσουμε ε, σταθερές δομές ενός μοντέρνου κράτους, να φτιάξουμε μια μοντέρνα IT. Βεβαίως, αυτό στην πραγματικότητα μπορεί να το κάνουν μόνο οι Αιτινοί. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε ο ΙΕ, ούτε οι δωρητές, ούτε ο ΙΕ, ούτε οι Αμερικάνοι μπορούν να το κάνουν. Ούτε μπορούν να κυδαιμονεύσουν αυτή τη χώρα Και ούτε μπορούμε να το φτιάξουμε ερήμην τους. Ούτε μπορούμε να φτιάξουμε ερήμην τους ένα μοντέρνο κράτος. Εκεί έγκυται η μεγαλύτερη δυσκολία, κατά την άποψή μου. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Προφανώς όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα και οι αιτινοί συνομιλητές μου το ίδιο θέλουν. Φυσικά χρειάζεται να ανοικοδομήσουμε τη χώρα. Παρ' όλα αυτά, ευκαιρία τώρα είναι να φτιάξουμε κράτος αιτινό. Αυτό τι σημαίνει. Καταρχήν, ότι οι δωρητές, παρότι δεν μου αρέσει πολύ αυτός ο όρος, δεν μου πολύ αρέσει αυτός ο όρος, έτσι. Θα πρέπει οι δωρητές πάντως να επιδείξουν επαρκή εξυπνάδα, γενεοδορία και δημοκρατικότητα για να αφήσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο πραγματικά όμως στους Αιτινούς. Γιατί αυτή τη φράση ότι οι πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι Αιτινοί το λένε όλοι. Έχει γίνει μπανάλ. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα γίνει αυτό στην πραγματικότητα. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος να γίνει, να υλοποιηθεί, να γίνει ο κανόνας και οι υπόλοιποι εμείς να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια χωρίς να παρεμβαίνουμε. Δεν είναι δουλειά δική μας να παρέμβουμε. Η δουλειά δική μας είναι να υποστηρίξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι ίδιοι οι Αιτινοί, που πρέπει να κάνουν για να φτιάξουν ένα μοντέρνο κράτος. Παράλληλα, ανοικοδομώντας βέβαια και τις υποδομές του, τη γεωργία του, και να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αυτή είναι η απόψή μου. Και αυτή είναι η δυσκολία που βλέπω. Επίσης ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει πραγματική κοινωνία των πολιτών. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα και σε άλλες χώρες. Δεν υπάρχουν πραγματικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Υπάρχουν στην πραγματικότητα θυγατρικές των ευρωπαϊκών ή αμερικανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων επιτόπου. Δεν υπάρχουν πραγματικές αυθεντικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και μέσα σε αυτή τη γενική φτώχεια που υπάρχει στην ΑΕΤ του πληθυσμού, αυτά τα στελέχη αυτών των θηγατρικών, τελικά αυτά τα άτομα θα γίνουν άτομα που θα έχουν το δεκαπλάσιο πούμε, του εισοδήματο του μέσου αιτινού. Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να το αφήσουμε να γίνει. Θα ήταν κακό για την κοινωνία. Επομένως, η ευθύνη μας είναι να βοηθήσουμε τους αιτινούς Πέρα από όλα αυτά, τώρα θα ήθελα να κάνω και ένα συγκεκριμένο ερώτημα που με ενδιαφέρει τα μάλα. Ερώτηση προς τον Δήμαρχο του Πογοπχάνς. Πώς επιλύουν το πρόβλημα της αποχέτευσης Υπάρχουν περισσότεροι Υπάρχουν περισσότεροι κουβανοί γιατροί, 700 τον αριθμό, από όλους τους υπόλοιπους γιατρούς μαζί. Πώς θα επιλύσουν το τεράστιο α, υγειονομικό πρόβλημα. Πώς το αντιμετωπίζουν λοιπόν το τεράστιο αυτό ε, πρόβλημα με την υγεία. Η κυρία Κρετή παρακαλώ. Θα μιλήσω ρουμανικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, διάφορες παρουσιάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την παρουσία της ε, σήμερα και για τη συζήτηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο του Πόχο Πχάνς για την παρουσία του καθώς και την κυρία Κολάχ Ε, θα ήθελα αρχίζοντας να μιλήσω για την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που έχει δύο σκέλη, την άμεση ανταπόκριση αλλά και την μακροπρόθεσμη προοπτική για την αναβάθμιση της χώρας, ε, της υγειονομικής κατάστασης, Ακούσαμε και τον συνάδελφο ε, Μαρτίνες ε, να εκθέτει το πρόβλημα. Πιστεύω και συνεχίζει αγγλιστή η κυρία Κρέτη ότι σε συνεργασία με τον κύριο Πίμπαλξ θα μπορέσετε να βρείτε μία λύση γιατί μετά από ε, τις ε, θερμό αντιδράσεις των πρώτων μηνών θα πρέπει να κάνουμε μακροπρόθεσμα πρόθεσμες προσπάθειες ε, για να υπάρχουν καλές οικονομικές και κοινωνικές ε, συνθήκες ε, για όλους και μην ξεχνάμε και τα παιδιά. Δυστυχώς πολλά έχουν μείνει ορφανά ή έχουν βρεθεί μακριά από τους γονείς τους. Υπάρχει εμπορία παιδιών, τέτοιου, απαγωγές παιδιών, τέτοιου είδους πράγματα ε, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θα ακούσουμε τον Δήμαρχο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πριν απαντήσω σε ερωτήσεις, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο για μία από τις υπόλοιπες παρουσιάσεις που ακούσαμε. Δεν θέλω τώρα να ε, δημιουργήσω πρόβλημα. Αλλά ήθελα να πω κάτι που ακούσαμε για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, στην ΑΕΤ. Ακούστηκε ότι δραστηριοποιείται κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, στο Πόχτο Πχάνς. Κανείς όμως δεν έρχεται να ζητήσει άδεια παρέμβασης στη διοικητική αρχή του ΠΟΓΟΠΧΑΣ Και άρα ε, δεν υπάρχει έλεγχος και γι' αυτό το λόγο στη δικιά μου την παρέμβαση σας ε, ανέφερα συγκεκριμένα ότι υπάρχουν σοβαρές επικαλύψεις των δράσεων. Και σε μία παρουσίαση Ακούστηκε επίκριση για την υπόθεση διφωνσή στο Πόχτο Πχάσε. Ε, μας μίλησε λοιπόν για την υπόθεση της Αγία ε, Ιδιοκτησίας. Ε, έχουμε εμείς ε, αρμόδια υπηρεσία, αλλά μην ξεχνάτε ότι ε, στο πόχτο πράσε κατά 80% δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας. Ε, δηλαδή ε, υπάρχουν παράνομες καταλήψεις σπιτιών. Δεν λειτουργεί κτηματολόγιο στο πόχτο πράσε. Γι' αυτό έχουμε τέτοιο πρόβλημα με τις ε, κοινωνικές υποδομές και γι' αυτό εγώ αγωνίζομαι ώστε στο πόχτο Πχάσε να υπάρξει να γίνει μια καταγραφή ούτως ώστε να καλύψουμε αυτή την έλλειψη του κτηματολογίου κατά την ανοικοδόμηση ε, της ΑΕΤΗΣ. Μιλήσατε για τη διάσκεψη στη Νέα Υόρκη, για την μικρή πρόοδο που σημειώθηκε, αλλά δεν επαρκεί αυτό διότι εάν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα είναι αδύνατο να γίνουν δημόσιες επενδύσεις ε, από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό. Είναι σοβαρότατο το πρόβλημα και οπωσδήποτε ε, θα πρέπει να παρέμβει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να λυθεί αυτό το θέμα. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω για τα, γενικότερα για τα προβλήματα ανοικοδόμησης ε, της ΑΕΤΙΣ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος και τις προτεραιότητες κατά την ανοικοδόμηση. Έκανα μία έρευνα ε, για το τι συνέβη στη Βηρητό, παραδείγματος χάρη. Ε, και η Βηρητός ε, κατεστράφη και υπήρξε βοήθεια, αλλά υπήρχε και μια υποδομή που ε, συγκροτήθηκε επί τόπου και υπήρχε κοινωνική αλληλεγγύη. Αλλά αυτή επέτρεψε να λυθεί το πρόβλημα του κτηματολογίου. Να ξέρουμε κάθε φορολογούμενος, κάθε πολίτης, ποιο κομμάτι γης είχε πριν την καταστροφή, οπότε μπορούμε κατόπιν προγράμματος να του προτείνουμε ένα άλλο αγροτεμάχιο, να του εξηγήσουμε πώς μπορεί να το αξιοποιήσει. Για να ε, τελεσφορήσουν οι προσπάθειές μου, σας το ανέφερα στην παρουσίασή μου, επέμεινα να υπάρξει καταγραφή της γης ε, και ζητούμε ε, βοήθεια στο Πόχτο Πχάς, για να έχουμε πόρους βιώσιμης ανάπτυξης για να μπορέσουμε να έχουμε και τον κατάλληλο προγραμματισμό. Είτε μιλάμε για την πολεοδομία, για την, γενικότερα για την ανοικοδόμηση, για την ανασυγκρότηση της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό είναι απαραίτητο κάποιοι. Μίλησαν για το σεισμό έκαναν ένα παραλληλισμό ανάμεσα στο σεισμό της Αιτής και το σεισμό της Χιλής. Ναι, αλλά με, στη Χιλή υπάρχει αυτή η βούληση συνύπαρξης και έτσι κατόρθωσαν να έχουν εφεδρικά σχέδια, έτσι κατάφεραν να ενημερώσουν ε, τους πολίτες ε, για τις φυσικές ε, καταστροφές. Πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Χρειάζεται μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που επικουρεί την ε, διοικητική αρχή και τους ερετούς αντιπροσώπους του λαού, τόσο ώστε να έχουμε ένα συνολικό σχέδιο για το Πόγο ε, δηλαδή πού θα οικοδομήσουμε, προς τα πού, πού θα εγκατασταθεί ο πληθυσμός κτλ. Κάτι άλλο που ανέφερε και ίσως σας σοκάρω τώρα αλλά πάντως το έγγραφο που παρουσιάστηκε στην ε, διάσκεψη της Νέας Υόρκη το διάβασα στην ιστοσελίδα. Δεν υπήρξε καμία ε, διαβούλευση για να συνταχθεί η δήλωση της διάσκεψης της Νέας Υόρκη. Πώς γίνεται αφού είμαι δήμαρχος του Πόχτο Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης είπε ένας ε, ότι είναι υπόθεση της ΑΕΤ η ανοικοδόμηση της ΑΕΤ ε, κατά προτεραιότητα. Ε, θέλουμε στη δική μου την πόλη να προετοιμάσουμε μια πρόταση ούτω ώστε ε, το Πόρτο Πράνς να συμμετάσχει στο εθνικό σχέδιο ανοικοδόμησης. Και για να κλείσω διότι ε, πήρα διάφορε σημειώσει από από τις ε, παρεμβάσεις Κύριε Μαρτίνες, ε, και εγώ ανατριχιάζω όταν ακούω τον όρο δωρητές. Καλό θα ήταν να μιλούσαμε για εταίρους και όχι για δωρητές. Ε, ως προς το υγειονομικό πρόβλημα τώρα, από το 1999 μέχρι το 2007 δεν είχε δήμαρχο Είχαμε ε, το Πορτοπράνς, είχαμε μία μόνο κεντρική εθνική αρχή και ξέρετε αυτό οδήγησε σε ε, μία ε, παρεμβολή των ε, κρατικών αρχών στις διοικητικές δομές των Δήμων και μέχρι στιγμής το 80% το κατήχε η Κεντρική Αρχή, δεν είχαμε αστυνομία. Πώς να χειριστούμε το θέμα της αποχέτευσης, το υγειονομικό πρόβλημα και ξέρετε οι κουβανοί οι γιατροί ήρθαν στο Δημαρχείο σε εμά να απευθυνθούν και σας διαβεβαιώ ότι εργάζονται με εξαιρετικό τρόπο. Και ξαναλέω ότι πρέπει τον Αιτιανό να ανοικοδομήσουμε ε, πριν από την Αιτή. Κάποιο που έχει χάσει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τι να του πούμε ότι, αρχίζουμε, ότι θα έχει σπίτι σε 15 χρόνια τώρα αρχίζουμε να χτίζουμε ένα καινούριο χωριό και με αυτό το χωριό, δηλαδή θα ξεπεράσει το δράμα, την τραγωδία του ε, με την ελπίδα αυτού του χωριού Χρειαζόμαστε χρόνο, περίσκεψη δεν θα σας υπαγορεύσω εγώ τι θα κάνετε βέβαια γιατί δεν είμαι και συνηθισμένο σε τέτοιου είδου κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις. Ήθελα μόνο να σας πω ότι ανησυχούμε πάρα πολύ και εγώ με την ιδιότητα του Γενικού Συντονιστή των Δημαρχείων της Μητροπολιτικής Περιοχής. Ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ ε, για τη συνεργασία μας και θα Θέλαμε να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει, ε, να οικοδομηθεί αυτό το κέντρο, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει πρόγραμμα του Πόγο Πχάνσε, η συμβολή του δηλαδή στο Εθνικό Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανοικοδόμησης. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ. Ε, σας καθησυχάζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία που μας κοινοποιείτε και τα εκτιμούμε ιδιαίτερα. Η κυρία Κρυσταλίνα Τζόρτζεβα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και χρήσιμη για όλους μας. Επιβεβαιωθήκαμε νομίζω σε κάποια από τα μηνύματα που είχαμε ακούσει και εμείς και κάποιες από τις πεπιθήσεις μας για τα νέα προβλήματα. Για μένα ήταν καινούριο αυτό που άκουσα ότι δεν ρωτήσαν τους δημάρχους για το σχέδιο ανοικοδόμησης. Ελπίζω ε, όταν αυτό αφορά τους Δήμους τους ε, να τους ρωτήσουν άλλη μόνο γιατί χωρίς ε, τοπική συμμετοχή συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν νοείται βιώσιμη ανάπτυξη στην ΑΕΤ. Επιτρέψτε μου να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που άμεσα ή έμεσα ετέθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το εγχειρίδιο της Παγκόσμιας Τράπεζας ε, για την ανοικοδόμηση. Ζήτησα από τους πρώην συναδέλφους μου να μου το στείλουν και το έπραξαν. Ε, είναι μια πλατφόρμα, μια πρόταση για όλους εκείνους που εργάζονται στην ΑΕΤ αυτό το καιρό και ε, ελπίζουμε να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση. Τώρα, για τις κοινότητες ε, που θα πρέπει να συνενωθούν και πάλι να ε, ζουν μαζί. Αυτά θα τα γνωρίζει καλύτερα από μένα ο Δήμαρχος. Αλλά εγώ τι είδα στην ΑΕΤ. Ακριβώς σε πολλές περιπτώσεις ε, γείτονε που έχασαν τα σπίτια τους γιατί καταστράφηκαν όλα μαζί μετακόμισαν όλοι μαζί στον ίδιο ε, καταβλισμό. Και διατηρείται έτσι ο κοινωνικός ιστός, δεν διανυγνύεται και μπορεί να βοηθήσει αυτό στην ανοικοδόμηση από κάτω προς τα πάνω. Ένα μικρό στρατόπεδο ή ένα τμήμα ενός καταβλισμού κάθε φορά. Ε, και αυτοί οι καταβλισμοί είναι σε περιοχές που πλημμυρίζουν και κινδυνεύουν από πλημμύρες και θα πρέπει να φύγουν. Είναι 30-35 χιλιάδες άνθρωποι που κινδυνεύουν πιο άμεσα από τους άλλους. Και τίθεται τώρα το εξής ερώτημα τους προσφέρει κάποια έκταση, οικόπεδα ε, η κυβέρνηση, αλλά είναι πολύ μακριά και αυτός είναι ένας δεύτερος ξεριζωμός. Είναι ένα δεύτερο δράμα, μια τραγωδία. Αυτοί έστω εγκαταστάθηκαν σε ένα καταβλισμό μαζί με κάποιους γειτονέ τους, ε, με ε, κάποια αντίσκηνα ε, και με τα στοιχειώδη προσπαθούν τώρα να φτιάξουν ένα καινούριο σπιτικό και πάλι τους διώχνουν. ή τους λένε επιτρέψτε στα σπίτια σας γιατί τα σπίτια σας είναι εντάξει, είναι ασφαλή. Ε, τώρα ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Από τη μια αυτό είναι κατανοητό από την ανθρώπινη σκοπιά, αλλά εκεί είναι που είναι ε, σε επικίνδυνες περιοχές, αυτό μπορεί να είναι και απειλή για τη ζωή τους την ίδια αυτή η αντίσταση του να φύγουν από εκεί. Αυτό μας λένε και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Αλλά ε, αυτό που μας ενδιαφέρει και πάλι είναι όσο γίνεται να ε, είναι σεβαστό αυτό το πνεύμα, το, συλλογικό, το κοινοτικό το, της ε, συνύπαρξης των γειτόνων. Τώρα, η προσέγγιση που αφορά το νησί ολόκληρο. Ε, Τώρα αισθάνομαι άβολα να τα λέω αυτά μπροστά στον Δήμαρχο, αλλά πήγα και στη Δομινικανή Δημοκρατία και το συζήτησα με τις αρχές εκεί. Και τι κατάλαβα εγώ, μετά από δεκαετίες ε, σχέσεων που ήταν δύσκολες και περίπλοκες μεταξύ γειτόνων, ε, βοηθάει η Δομινικανή Δημοκρατία. Ήταν η πρώτη υπηρεσία πολιτικής προστασίας που πήγε να βοηθήσει για τη διάσωση των Αιτινών. Και επίσης πολύ μεγάλη υποστήριξη για τα αποθεματικά, για τα υλικά, για την επιμελητία και την υποστήριξή τους. Και βοήθησε τριπλά την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Ε, δεν θα πρέπει να λησμονούμε και τη ικανή δημοκρατία όταν θέλουμε βοήθεια. Δηλαδή την αποκατάσταση των αποθεμάτων, την ανανέωσή τους, γιατί τώρα επίκενται κυκλώνες ε, και μάλιστα πιο ισχυρή από το μεσόρο. Και αυτοί θα πλήξουν όλο το νησί, και την ΑΕΤ και τη Δομικανή Δημοκρατία. Αν λοιπόν τα αποθέματα τη Δομικανή Δημοκρατία εξαντλούνται, διακυβεύεται αυτή η ε, εύθραυστη αδελφοσύνη που έχει πλέον προκύψει από την ε, τραγωδία και μετά θα τρέχουμε να σώσουμε και την άλλη χώρα. Και ε, τα προγράμματα είναι προγράμματα συνεργασίας και κατέρωθαν για το πώς μπορούν να συνεργάζονται οι δύο χώρες και στην πολιτική προστασία και παντού. Η ΑΕΤ τώρα ε, επιθυμεί έτσι, πολύ πιο έντονα να ε, αποκτήσει δομές αντιμετώπισης αλλά και πρόληψης κυρίως των κρίσεων και, και τις Και με ένα πραγματικό εταίρο που είναι ο γείτονά του ο άμεσος. Αξίζει να υποστηριχθεί αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα για ε, τη Μεθόριο. Μαθαίνουμε ότι ο κόσμος έφυγε από, τα, από την παραμεθόριο περιοχή για να πάει στη δομικανή δημοκρατία για να ζήσει με συγγενείς του, με γνωστούς, με φίλους και αυτό ε, ενδεχομένω ε, θεωρείται κίνδυνος μεταναστευτικό ρεύμα. Βεβαίως όσο περισσότερα κάνουμε εμείς για να υποστηρίξουμε και για την απασχόληση και να ανακουφίσουμε την ανθρωπιστική κρίση τόσο λιγότερη θα είναι η μετανάστευση προς τη δομικανή δημοκρατία και λιγότερη η πίεση στις σχέσεις ε, των δύο χωρών που κινδυνεύουν από καλές που είναι τώρα ξανά επιδεινωθούν. Τώρα, ε, τι κάνουμε με το γεγονός ότι είναι περιορισμένες, ε, όπως και να έχει το πράγμα, οι δομές και οι θεσμοί στην ΑΕΤ. Η αποκέντρωση πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίσιμη και με τη διπλή έννοια. Ε, ελπίζω να μην διαφωνήσει πολύ ο Προδήμαρχος. Αυτό σημαίνει να δημιουργηθούν δραστηριότητες, κέντρα αναπτυξιακά εκτός της πρωτεύουσας, εκτός του Port-au-Prince. οχι ε, για να μειωθεί η σημασία του Port-au-Prince, αλλα για να είναι ένας πιο ε, βιώσιμος από ό,τι είναι σήμερα. Και αποκέντρωση επίσης με την έννοια της εκχώρησης αρμοδιοτήτων. Ε, μου έκανε εντύπωση αυτό που είδα ότι ακόμα και σε τέτοια καταστροφή λειτουργούσαν κάποια πράγματα. Ε, όπου ήταν αρμόδια η τοπική αυτοδιοίκηση και ενεργή και όπου ήταν ε, πραγματικά ε, επαγγελματική διαχείριση και των καταβλισμών. Υπάρχουν πολλοί λοιπόν στην ΑΕΤ και χάρηκα γι' αυτό που μπορούσαν να ηγηθούν των τοπικών κοινοτήτων. Είδα μέρη όπου ε, ήταν διορισμένοι δάσκαλοι χωρίς να ήταν δάσκαλοι. Και μας έλεγαν οι ντόπιοι και οι θυνοντές ότι τα παιδιά μας δεν πάνε στο σχολείο μήνες ολόκληρους, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Διότι πάνε, παίρνουν κάποιον, το διορίζουν εδώ λοιπόν, εσύ τώρα θα είσαι δάσκαλος. Ε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να, να υφανθεί αυτός ο κοινωνικός ιστός με ε, πολύ μικρά τοπικά έργα που να ενεργοποιούν και να δραστηριοποιούν αυτό το πνεύμα της τοπικής συνεργασίας και των τοπικών κοινοτήτων. Και ένα τελευταίο, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς ενέχεται σε αυτά. Εγώ θα μιλήσω εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 580 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι ε, 120 εκατομμύρια για την ανθρωπιστική βοήθεια και 460 για την αναπτυξιακή. Εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις. Ε, ολοκληρωμένα δίνουμε αυτή τη βοήθεια και την ανθρωπιστική και την ε, αναπτυξιακή. Είναι λένδετα και το ένα οδηγεί στο άλλο. Κάποιο είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, ε να βοηθούμε τον κόσμο, τα σημαντικότερα είναι η παιδεία, η υγεία και η απασχόληση. Για να έχει ο κόσμος μια πρώτη ελπίδα ε, στην IT. Και αυτό σημαίνει ότι όποιο έργο και να κάνουμε, όποιο project στην υποδομές στη γεωργία, θα πρέπει να βάζει στο επίγεντρο της προσοχής του τον άνθρωπο. Ας σταματήσω καλύτερα εδώ. Κάποιος είπε ότι θα παραμείνουμε εκεί. Βεβαίως και θα παραμείνουμε. Μετά την εποχή των κυκλώνων θα πάω στην ΑΕΤ γιατί μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση και οι ανάγκες οι ανθρωπιστικές για να δούμε ε, τι χρειάζεται να κάνουμε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Παραμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επειδή είναι τεράστιο το έργο αλλά και πολύ μεγάλη η γενεοδορία των ανθρώπων και νομίζω ότι θα παραμείνουμε εκεί για να δούμε τι πρέπει να κάνει, πώς να βοηθήσουμε. Ο κόσμος το περιμένει αυτό από μας. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Madame Commissaire. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Άλλε παρεμβάσει, ε, άλλες ερωτήσεις. Αν όχι, θα πάμε στο επόμενο σημείο, σημείο 8. Δεν υπάρχουν ερωτήσει. Θα μιλήσουμε τώρα για την αποτελεσματικότητα τη αναπτυξιακή βοήθεια με τον κύριο Καλτερίζη, που έχει γράψει το βιβλίο ε, Η Αφρική μπορεί να βγει από τη δυσκολία τη. Γιατί η ξένη βοήθεια δεν δίνει αποτελέσματα. Τώρα σε πριν από λίγα χρόνια ε, είναι τώρα υπάλληλο στην ε, Διεθνή Τράπεζα και είναι εμπειρογνώμονα εδώ και πάνω από 30 χρόνια για αυτά τα θέματα. Γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα των αναπτυσσόμενων χωρών. Ε, το σκλαβοπάζαρο, η απεικιοκρατία, η παγκοσμιοποίηση δεν είναι αυτή η ένοχη. για την σημερινή κατάσταση της Αφρικής για τα προβλήματα άλλων περιοχών του κόσμου, αλλά η διατήρηση δικτατορικών καθεστώτων που είναι διεφθαρμένες και που στηρίζονται και από την ξένη βοήθεια. Θα συζητήσουμε για την άποψή σας για αυτό το θέμα και κυρίως για τις προτάσεις για να βοηθήσουμε πραγματικά τις αναπτυσσόμενες χώρες. Κύριε Καλντερίζη, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ. ακούτε? Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ε, μεγάλη μου τιμή που με προσκαλέσατε στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα να πω από την αρχή ότι όταν μιλάμε για βοήθεια, δεν θα μιλήσω, δεν μιλάω για την ανθρωπιστική βοήθεια και την ε, ανακούφιση των κρίσεων. Δεν πιστεύω ότι οι φτωχοί και οι άρρωστοι θα πρέπει να υποφέρουν γιατί είναι, διευθύνονται από διεθαρμένες ε, κυβερνήσεις. Εγώ μιλάω για την κλασική βοήθεια που πηγαίνει στι αναπτυσσόμενες χώρες, τους ε, προϋπολογισμούς τους, ε, από τις πλούσιες χώρες. Οι επικρίσεις μου για την ξένη βοήθεια οικοδομούνται γύρω από τον άξονα της ε, κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτές είναι οι προσωπικές μου απόψεις και στον Καναδά ψηφίζω σοσιαλιστές και πράσινους. Βλέπετε αυτές είναι οι απόψεις μου. Όταν ονειρεύομαι για μια καλύτερη Αφρική, μια καλύτερη Αφρική, και πρέπει να σας πω ότι 30 χρόνια ασχολήθηκα με την Ήπειρο αυτή, είχα, η πιο ενδιαφέρουσα συνάντηση που είχα ήταν με μία νοσοκόμα ε, στην, σε μία πόλη στο Côte d'Ivoire, ε, στη Δυτική Αφρική. Ένα πρωί προσπαθούσα να καταλάβω αν τα εκατομμύρια ε, δολαρίων που στέλνουν οι δυτικοί στην Αφρική έχουν αποτέλεσμα. Το αποθαρρυντικό είναι ότι πήγα και είδα άδεια νοσοκομεία, χωρίς να υπάρχει βασικός εξοπλισμός, χωρίς να υπάρχει νόπνευμα, ε, χωρίς να υπάρχουν στρώματα, χωρίς να υπάρχουν γάζες, ε, χωρίς να υπάρχουν ε, σεντόνια, ε, σε, μια, σε ένα γυναικολογικό τμήμα ενός νοσοκομείου, μια γυναίκα ισχυστεί κατά τη διάρκεια της γένας και η μέα που έπρεπε να τη ράψει, χρειάστηκε να τη ράψει με χάλκινο σύρμα. Ήταν το μόνο πράγμα το οποίο υπήρχε στη διάθεση της. Πήγα και σε μια άλλη κλινική. Συνάντησα μια νεαρή νοσοκόμα. Εκεί είχε όλο ο χρειαζόταν. Uh, uh, να Στο Αμπιτζάν. Ε, είχε όλα τα περίεργα ιατρικά πράγματα, αλλά δεν είχε νερό. Και διαρωτώ γιατί αυτή η διαφορά. Ε, στην πραγματικότητα ε, ζητούσε βοήθεια από τον κόσμο. Ε, το κράτος δεν βοηθούσε. Χάρη στην εξυπνάδα της και στις έντεχνες λύσεις που έβρισκε, πραγματικά έβρισκε λύσεις. Ε, ήταν επικεφαλής, είναι επικεφαλής ε, τώρα εδώ και 11 χρόνια αυτής της κλινικής και τα πάει πάρα πολύ καλά. Ε, αυτό εκεί στην περιοχή λέγεται κοινωνική επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ε, άνθρωποι στον αναπτυσσόμενο κόσμο όπου πραγματικά θα έπρεπε να είναι αποδέκτες της οικονομικής βοήθειας από τη Δύση. Ένα μεγάλο πρόβλημα με τη βοήθεια είναι ότι δεν είναι αρκετά σημαντική. Ε, επίσης σημαντικό είναι η, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι σωστές ε, πολιτικές από την κυβέρνηση, η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη. Την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των φτωχών στον κόσμο, όσοι ζουν με λιγότερα από 2 δολάρια τη μέρα, μειώθηκε κατά 9%. 200 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αυτοί. Ε, και αυτό, αυτή η μειωσία έγινε χάρη στην βελτίωση στη γεωργία. Η γεωργία ε, πρέπει να είναι ο βασικός στόχος των ε, πολιτικών των κυβερνήσεων στην Αφρική. Αλλά δυστυχώς ε, υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις εναντίον της γεωργίας στην πραγματικότητα, αν διορθώσουμε αυτή την προκατάληψη, νομίζω θα άρουμε πολλά εμπόδια που βαραίνουν τον ε, Γεωργό. Η βοήθεια μπορεί να τον... Η απτυξιακή βοήθεια μπορεί να τον βοηθήσει. Αλλά το βασικό θα ήταν να έρθουν τα εμπόδια προς τους γεωργούς. Ε, γιατί οι κυβερνήσεις δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Η εξωτερική βοήθεια όμω μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά απλώ θα πρέπει να χρησιμοποιείται διαφορετικά. Από την πείρα μα βλέπουμε ότι η βοήθεια είναι αποτελεσματική μόνο στις χώρες όπου οι κυβερνήσεις τους προωθούν την ανάπτυξη και την καλύτερη διανομή του εισοδήματο ε, μέσω πολιτικών, ε, επενδύσεων ε, και σοβαρών προσπαθειών. Η βοήθεια δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για φακελάκια, για προμήθειες, ή να καλύψει ας πούμε, την αδιαφορία των, των κυβερνήσεων που δεν ασχολούνται με την ανάπτυξη. Πολύ λίγοι είναι υπέρ της ξένη ξένης βοήθειας. Οι κυβερνήσεις ε, δεν ξέρουν, οι τόπιες κυβερνήσεις δηλαδή, δεν ξέρουν πώς να τη χρησιμοποιήσουν, το χρησιμο... τη θεωρούν σαν αναγκαίο κακό. Ούτε οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις αρέσκονται στην ξένη βοήθεια γιατί πιστεύουν ότι είναι σε ανταγωνισμό με τους δικούς τους προϋπολογισμούς. Ακόμη και οι υπάλληλοι που ασχολούνται με την ε, ξένη βοήθεια δεν είναι πολύ θερμοί. Γιατί αισθάνονται ότι δεν μπορούν να φτάσουν στους πραγματικούς στοχούς. Ε, οι δυτικοί που πιστεύουν στην ε, κοινωνική δικαιοσύνη και οι μεταρρυθμιστές στην Αφρική που πιστεύουν ότι η βοήθεια ε, στην πραγματικότητα ενισχύει τους, ε, τις αυταρχικές κυβερνήσεις, ε, δεν πιστεύουν. Δεν πιστεύουν στην βοήθεια. Θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα για να πιστέψουν και αυτοί. Ε, ξέρω ένα ε, κάτι πρόσφυγες πρόσφυγες από το Σουδάν που ζουν τώρα στον Καναδά, στη βορειοδυτική, στο βορειοδυτικό τμήμα του Καναδά. Ένα πρωί ξύπνησαν και βρήκαν μπροστά στον κήπο τους ε, βρήκαν μπροστά τους ένα αποκεφαλισμένο κεφάλι ζώου. στην πραγματικότητα ήταν ένα έθιμο της χώρας τους, ε, ένα είδος βοήθειας. Αλλά μοιάζει η εξωτερική βοήθεια σαν αυτό το αποκεφαλισμένο ε, ζώο. Ε, δεν μοιάζει καλή. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί, θα αρχίσει να μοιάζει πιο θετική μέχρι να χρησιμοποιηθεί πιο σωστά. Θέλω να πω κάτι ριζοσπαστικό εδώ. Γιατί να υπάρχουν 12 και 13 υπηρεσίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να ασχολούνται με την ξένη βοήθεια αντί για 2 ή 3. Ε, πολύ περισσότερα τμήματα της βοήθειας θα πρέπει να πηγαίνουν στο να βοηθήσουν παράλληλα πολλές χώρες ή όλη την ε, Ήπειρο για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων κατά της εφηματίωσης του AIDS και τα λοιπά, ε, Βοήθεια για τη γεωργία, ε, για την ανάπτυξη των πανεπιστημίων και το υπόλοιπο θα πρέπει να πηγαίνει σε συγκεκριμένες χώρες όπως η Γκάνα και η Μοζαμβίκη, οι οποίες έχουν δείξει εδώ και πολλά χρόνια ότι μπορούν να διαχειριστούν τους πόρους τους και την βοήθεια να τη διαχειριστούν αποτελεσματικά. Ίσως 10 από τις 48 υποσαχάριες ε, χώρες της Αφρικής ε, εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Οι υπόλοιπε χώρες ε, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν πιο σκληρούς όρους, διεθνή εποπτεία, παρατηρητές στις εκλογές τους, επιθεωρήσεις. Όταν ψηφίζονται σημαντικά προγράμματα στην Βουλή για τα δημοτικά ας πούμε κτλ. Ε, θα πρέπει τελικά το αποτέλεσμα να είναι η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Ε, αλλά αυτό θα γίνει μόνο με αυστηρότερους όρους. Η βοήθεια θα πρέπει να δίνεται με τρόπο πιο διαφανή και ορατό. Να υπάρχουν προϋποθέσεις πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέει τη δημοκρατία και την ανάπτυξη, ενώ οι άλλοι οι υπόλοιπε χώρε αδιαφορούν για αυτό το θέμα, για αυτή τη σχέση. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Δανία όμω και ο Καναδά λένε ότι η Αφρική είναι η πρώτη προτεραιότητα, αλλά ε, παρόλα αυτά δίνουν τα περισσότερα χρήματά του για την ξένη βοήθεια ενώ στο Αφγανιστάν. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, ο τρόπος ε, με τον οποίο η, μια κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους πολίτες, τους ε, μικρούς γεωργούς, τους ε, επιχειρηματίες, τους δημοσιογράφους, θα πρέπει να είναι προϋπόθεση για το επίπεδο της βοήθειας που λαμβάνει η χώρα. Έπειτα θα πρέπει να είναι ο κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο δίνεται και να εξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο το δίνουμε, τόσο ώστε και ο Αφρικανός, πέρα από τις κυβερνήσεις, να καταλαβαίνουν τι παίζεται. Νομίζω ότι Παραδείγματο χάρη, θα πρέπει να φτιάξουμε ε, αυτοκινητόδρομους, μεγάλους αυτοκινητόδρομους στην Αφρική και να ε, υπάρχει ένα πρόγραμμα ας πούμε, ε, συντήρησής τους, ε, παρά να τους ξαναφτιάχνουμε από την αρχή κάθε χρόνο. Επίσης, θα πρέπει η βοήθεια να συμπληρώνει τα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων, ούτως ώστε να μην υπάρχει έτσι διαρροή υπαλλήλων προς τη Δύση κτλ. Και έπειτα θα πρέπει στους στοχούς να συμπληρώνει το εισόδημά τους όπως παραδείγματο χάρη κάνουν οι κυβερνήσει στη Βραζιλία και σε άλλες χώρες, συμπληρώνουν το εισόδημα των φτωχών για να τους βοηθήσουν να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή, θα πρέπει να, ε, χωρίς να είμαστε πατερναλιστές, να παρακολουθούμε τα πράγματα ούτως ώστε οι στόχοι να υλοποιούνται. Μια άλλη αρχή επίσης θα πρέπει να είναι εξής, ότι οι κυβερνήσεις δεν θα έχουν δικαίωμα σε βοήθεια. Έχει νόημα α, μόνο να δίνεται ως επένδυση για το μέλλον. Συμπληρωματικά με αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Όχι οι κυβερνήσει αυτόματα να έχουν δικαίωμα σε βοήθεια. Επίσης οι αφρικανικές κυβερνήσεις. Ποια στάση θα πρέπει να έχουν. μπορεί να έχουν δικαίωμα να ζητήσουν περισσότερους πόρους εάν είναι αποτελεσματικοί στην χρήση. Με απλές διαδικασίες, ε, αποτελεσματικές και λογοδοσία εκ μέρους τους. Επίσης, θα πρέπει οι αφρικανικές κυβερνήσεις να μην δίνουν δουλειά σε ξένους, για μελέτες κτλ. Ε, είναι σημαντικό αυτό για μας, αλλά όχι για αυτούς. Ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια διασπάθηση χρήματος. Ευτυχώς κάποιες ε, φτωχές χώρες ε, σταματούν να το παίζουν θύματα και έχουν μια πιο έτσι, θετική στάση. Ο Παλ Καγκάμε, πρόεδρος Αφρικανικής Κυβέρνησης, που έχει τη συμπάθεια του κόσμου, 15 χρόνια μετά τη γενοκτονία, είπε κανένα δεν χρωστάει τίποτα στη Ρουάντα, είναι πρόεδρος του ε, Ρουάντα». Και ένας άλλος πρόεδρος είπε ότι οι Βρετανοί μέσα σε πέντε χρόνια ε, έφτιαξαν ένα συνδυρόδρομο από τις ε, ακτές της Κένιας μέχρι το εσωτερικό μέσα σε πέντε χρόνια η Κένια αύξησε τα φορολογικά της έσοδα τα τελευταία χρόνια γιατί μείωσε τις αθέμητες πρακτικές, τις άτιμες πρακτικές, τη διαφθορά, ε, στην εφορία της. Και το έκανε γιατί. Γιατί λάβανε πολύ μικρή βοήθεια, 5% η Κένια σε σχέση με το 40% που παίρνει Τανζανία και η Ουγγάντα αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα με τις, ε, με τις κακές επιπτώσεις μερικές φορές ε, της βοήθειας. Αλλά και δείχνει πόσο σημαντικό είναι η ατομική πρωτοβουλία, όπως αυτή που ανέφερα στην αρχή της νεαρής ε, νοσοκόμας. Σας ευχαριστούμε. Τώρα θα αρχίσει η ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής μας. Ποιος θα ήθελε παρακαλώ το λόγο. Ο κύριος Μίτσελ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ομιλητή. Ε, βρήκα ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο του, κύριο Καλντερίση. Φοβούμαι ότι αν αρχίσουμε να λέμε σε όλους ότι δεν βοηθάει η βοήθεια, θα βρούνε καλό λόγο για να μην φτάσει στο 0,7% το ποσοστό που πρέπει. Δηλαδή να δώσουν ναι, για ανθρωπιστική βοήθεια και μπορεί να μην φτάσει ποτέ η βοήθεια στις χώρες που τη χρειάζονται. Γι' αυτό και δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω Ξέρω, η World Vision έχει αντίθετη άποψη. Λέει ότι ε, είναι αποτελεσματική η διεθνής βοήθεια. Ε, γνωρίζω κάποια από τα παραδείγματα του κυρίου Καλντερίζη και γνωρίζω τις προσωπικές του εμπειρίες. Αν πούμε ότι πολλές με κυβερνητικέ οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Αφρική και σκεφτείτε τώρα μια χώρα σαν τη δική μου, ε, πάνε οι Ιρλανδοί στην Αφρική και προσπαθούν να φτιάξουν σπίτια εκεί. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ε, εμείς το 70 παραδείγματος χάρη ιδιωτικοποιήσαμε οικοδομικά συγκροτήματα ε, και δεν τα είχε η κοινότητα και δυσκολεύτηκαν κάποιοι να, καταλάβουν ότι είναι πλέον ιδιοκτήτες. Τι εννοώ. Μήπως είναι υπερβολικό να λέει κανείς ότι δεν είναι αποτελεσματική η βοήθεια. Αν δεν, δεν είναι αποτελεσματική η βοήθεια, τι, τι μπορεί να βοηθήσει λοιπόν για να βελτιωθεί η κατάσταση και πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο 0,7% του προϋπολογισμού που πρέπει να διοχετεύεται στη βοήθεια. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ ε, και μας κάνετε να ε, σκεφτόμαστε, αλλά α κάνω και εγώ να σκεφτείτε. Χριστιανοδημοκράτε πρέπει να ψηφίζετε, όχι πράσινου ε, και σοσιαλιστέ ε, στον Καναδά. Οπότε αυτό που σα ανέφερα, τι, ε, πώ το, σχολιάζετε, τι μπορεί να αντικαταστήσει τη βοήθεια. Ευχαριστώ, κυρία Λεβίνα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καλτερίζη. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή του. Δυστυχώ εγώ δεν το διάβασα το βίβλιο σας, αλλά έχω διαβάσει εσχάτω άλλα. Dead Aid και ένα του Αγκάρι Ματάι, μια πρόκληση για την Αφρική τιτλοφορείται. Πήρε το, πριν από δύο χρόνια το Νόμπελ Ειρήνης, είναι κενιά Μετά λοιπόν από την ανάγνωση αυτών των βιβλίων ε, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα. Δηλαδή ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποιος είναι ο ουσιαστικός αντίκτυπος ε, της βοήθειας ε, σε πολλές υποσαχάριες αφρικανικές χώρες. Η Ρογκάη Ματάη λέει στο βιβλίο της ότι έχει ε, και αρνητικό αντίκτυπο η βοήθεια σε πολλές ε, τέτοιες αφρικανικές χώρες ε, νοτίου της Σαχάρας. και ότι δεν είναι κανείς υπόλογος τελικά, δεν επομίζονται τις ευθύνες αυτοί που διαχειρίζονται την βοήθεια και ότι επιρρύπτεται η ευθύνη στους δωρητές. Αυτό δεν βοηθάει στην, στον εκδημοκρατισμό των καθεστώτων όταν δεν υπάρχει, δεν είναι κανείς υπόλογος. αν δεν ε, ε, δίνει κάποιος λογαριασμό στους ε, φορολογούμενους καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι εντελώς, γίνεται εντελώ αδιαφανής. Επίσης η διαχείριση της κρίσης, η οικοδόμηση των σχολείων, των νοσοκομείων, πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει απ' έξω να έρθει η βοήθεια στο βιβλίο του Μπίσα Μόγιος. Ε, ήταν αμφιλεγόμενο το βιβλίο, αφήστε που είναι ταμπού το θέμα, ότι δεν είναι απαραίτητα καλή η βοήθεια. Λοιπόν, πώς σχολιάζεται το συμπέρασμά της Συμφωνείτε ως προς την ανάλυση από ό,τι διαπίστωσα, αλλά πώς σχολιάζετε το συμπέρασμά για την πρόθεση του εμπορίου αντί για χορήγηση βοήθειας. Μιλήσατε επίσης για τις νέες αρχές που πρέπει να διέπουν την ε, χορήγηση βοήθειας. ποια είναι η καλύτερη μέθοδος που μπορούμε να, να ακολουθήσουμε. Κάτι άλλο που συζητείται στην γενέτειρά μου σε μεγάλο βαθμό είναι ότι πολλές φορές η βοήθεια μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της διαφθοράς. Πώς το σχολιάζετε. La parole est à Mme Keller. Ευχαριστώ κυρία Κέλλερ, έχει το λόγο τώρα. δηλαδή. Ευχαριστώ. Ε, Ούτε εγώ διάβασα το βιβλίο. Ε, ε Αφρική γιατί δεν αποδίδει η εξωτερική βοήθεια ε, ένα άλλο βιβλίο. Δηλαδή πώς μπορεί κανείς να κάνει μια καλή δουλειά που παρόλα αυτά να είναι μια τρύπα στο νερό. Και τι πρέπει να κάνουμε για να αποδίδει και αυτή η δουλειά μας. Μιλήσατε για τις εξωτερικές επενδύσεις, για τις ξένες επενδύσεις. Δεν είμαι βέβαιη ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έχουν δυνατότητα να προσελκύσουν και τόσο πολλές ξένες επενδύσεις. Επίσης είπατε ότι η βοήθεια ενδεχομένως να οδηγήσει σε ε, κάποια ανευθυνότητα των κυβερνήσεων, ακριβώς γιατί όταν είναι ξένες επενδύσεις δεν είναι υπόλογες κυβερνήσεις ή ηθήνοντες. Ε, ναι, αλλά τι είναι αυτό που κάνει μια κυβέρνηση να λογοδοτεί. Είναι η κοινωνία των πολιτών που χειραφετείται και απαιτεί να λογοδοτεί η κυβέρνηση όχι εμείς έξωθεν δηλαδή να επιβάλλουμε τέτοια πράγματα. Για, για να υπάρξει η κοινωνία των πολιτών στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες θέλουν υποστήριξη και οικονομική και Επίσης ένα ελεκτικό συνέδριο, δεν ξέρω, ένα, ένα σώμα ελεγκτών. Πώς θα το κάνετε αυτό, ποια, πού θα είναι οι πόροι. Με βοήθεια που δεν είναι πραγματικά ανεπτυξιακή βοήθεια, είναι μάλλον επικούρηση, ε, είναι χρήματα που εμείς έχουμε πάρει από τις χώρες αυτές και προσπαθούμε τουλάχιστον μέρη να τους τα επιστρέψουμε. Λοιπόν, ε, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ε, καταστούν υπόλογες, αλλά ακριβώς με ενίσχυση του πληθυσμού, της κοινωνίας των πολιτών, του λογιστικού ελέγχου και όλα αυτά με τρόπο υπεύθυνο για το πώς δαπανώνται τα χρήματα. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση που ακούσαμε, στέλνουμε επόπτες ας πούμε δωρητές. Δηλαδή άλλοι Ευρωπαίοι που να πάνε στην Ταζανία, ξέρω εγώ, και να ε, εποπτεύουν τι κάνει η κυβέρνηση της Ταζανίας ε, με τα χρήματα αυτά. Χρειάζεται ε, τοπική πίεση, δηλαδή από την ίδια την κοινωνία, την κοινωνία των πολιτών της χώρας. Και το θέμα της αναπτυξιακής βοήθειας δεν είναι μόνο ε, η λογοθεσία των ε, χωρών που δίνουν στα κοινοβουλιά τους και στη δική τους κοινή γνώμη. Αλλά οι αποδέκτριες χώρες θα πρέπει οι δικαιούχοι να αναπτυχθούν. Δεν μου αρέσει αυτό το θέμα της εποπτείας των δωρητών. Γιατί πολλές φορές και οι διορίτριες χώρες δεν θέλουν να φαίνεται και πάρα πολύ που πηγαίνουν τα χρήματα, γιατί έχουν και ίδιο συμφέρον να χρηματοδοτούν δικούς τους χώρες αυτές. Και πώς θα πηγαίνουν τα χρήματα τελικά στους πολιτές οικογένειες, είπατε. Υπάρχουν πολύ φτωχοί άνθρωποι ε, και το εισόδημά τους εξαρτάται από την αναπτυξιακή βοήθεια. Εκεί το άλλο θέμα το φορολογικό. Γιατί είναι και αυτό είναι τόσο μεγάλο ζήτημα, γιατί τις τελευταίες δεκαετίες εμείς, ο βοράς, οι αναπτυγμένοι, τι, τι λέγαμε στον κόσμο, μειώστε την κρατική ε, παρέμβαση, φίλε ελευθεροποιηθείτε, απελευθερώστε, αφήστε τους φόρους. Το θέμα δεν είναι ότι φταίνε πάντα οι αναπτυσσόμενες χώρες, κάτι πάει στραβά. Έχει πάει πολύ στραβά με τη δική μας ε, ε, αναπτυξιακή βοήθεια, με ρωτάτε και εμένα τη γνώμη μου. Μάλλον εκεί λοιπόν εστιάζεται περισσότερο το πρόβλημα και ήθελα να πω και κάτι άλλο, δεν το βρίσκω και το έχω ξεχάσει, αλλά δεν πειράζει. Να βελτιώσουμε λοιπόν την αναπτυξιακή μας βοήθεια με διαφορετικό τρόπο, να είναι και προβλέψιμη και με σαφήνεια. Βεβαίως συμφωνώ με το μορατόριο. Βέβαια είναι πολύ λίγα τα χρήματα τώρα, μπορεί να τους τα έχουμε ε, υποσχεθεί αλλά δεν τα έχουμε τα χρήματα όπω το 0,7%. Λοιπόν, μια συνεκτική προσέγγιση, όχι να τα δίνουμε με το ένα χέρι και με το άλλο να τα παίρνουμε πίσω και ε, να έχουμε και τα θετικά παραδείγματα. Λέτε ότι το πρόβλημα ποιο είναι με την Αφρική. Στην Αφρική βέβαια έχουμε πάντα προβλήματα, φασαρίες, βάσανα, χρήματα που χάνονται κτλ. Και η κυρία Μόγιο έδωσε ένα παράδειγμα θετικό, αλλά βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο βοήθησε η αναπτυξιακή βοήθεια γι' αυτό, αλλά δεν είναι όλα ε, στραβά. Και βέβαια οι στόχοι η για την χιλιετία δεν μπορούν ποτέ να εκπληρωθούν με τα τόσο λίγα χρήματα που δίνουμε σήμερα. Ο κύριος Μαρτίνες τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα είμαι αρκετά σύντομος. Πρώτον, διότι συμφωνώ με ε, τα όσα είπαν οι δύο προλαλήσασες. Εγώ θα είμαι πιο ομός ε, και σε σχέση με αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Γκέι Μίτσελ. Για να είμαι ειλικρινής, αυτός ο τίτλος του βιβλίου δεν με ενδιέφερε πάρα πολύ, αλλά με ανησυχούσε. Δηλαδή, ωραίος τίτλος είναι, αλλά ε, και λίγο προβοκατόρικος Ίσως έχω γεράσει εγώ πολύ για να μπορούν να με ε, προκαλούν με αυτά τα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει ο τίτλος. Ούτε είναι σαφής. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι η Αφρική και ε, what's the trouble with Africa και τι γίνεται με την εξωτερική βοήθεια. Δεν ξέρω, το foreign aid αυτό εννοείται, απτυξιακή βοήθεια. Τι θα πει εξωτερική βοήθεια. Ή μήπως είναι η βοήθεια στην εκμετάλλευση τι θα πει foreign aid ναι, εδώ γενικά και αόριστα, είναι απτυξιακή βοήθεια. Αν ναι, πρέπει να πω στον κύριο Καλτερίζη ότι καταρχάς μπορώ να σας πω εγώ, μισή σελίδα θέλω, δεν χρειάζομαι βιβλίο ολόκληρο, ορίστε μια σελίδα α5 για να σας πω <laughs> γιατί υπάρχει πρόβλημα στην Αφρική. Κοιτάξτε λοιπόν να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα στην Αφρική. Αυτά που τα χρήματα που δίνουμε για βοήθεια, που είναι πάρα πολύ λίγα, και από την άλλη τους τα παίρνουμε επί 100 έτσι αυτό είναι το πρόβλημα στην Αφρική. Το πρόβλημα δεν είναι εξωτερική βοήθεια. Το πρόβλημα είναι αυτό που τους παίρνουμε όταν τους δίνουμε ένα κλάσμα στην Αφρική και το πολλαπλασιάζουμε. Εντάξει, αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί. Πρώτον, αν αυτή η εξωτερική βοήθεια, μάλλον χωρίς αυτή τη βοήθεια, θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Στην καταπολέμηση του AIDS, στην καταπολέμηση ε, του αναλφαβητισμού και σε πολλά άλλα θέματα. Γιατί η εξωτερική βοήθεια δεν είναι μόνο η βοήθεια που φτάνει στην Αφρική από τις χορούλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Βόρειας Αμερική. Η εξωτερική βοήθεια τους φτάνει ας πούμε και από την Κούβα εκεί. Όπου αυτή τη στιγμή έχουμε 20.000 κουβανούς γιατρούς που δουλεύουν στην Αφρική. Και αυτό εξωτερική βοήθεια είναι. Κάθε μέρα θεραπεύουν αρρώστους. Γιατί η έλλειψη εξωτερική βοήθειας ακριβώς οδήγησε στο γεγονός να φεύγουν οι γιατροί του και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες όπου ε, είχαν υποτροφίες και σπούδασαν δικές μας από τον αναπτυγμένο μας ε, υποτίθεται κόσμο. Κοιτάξτε λοιπόν το πρόβλημα της Αφρικής δεν είναι εξωτερική βοήθεια. Η εξωτερική βοήθεια, η αναπτυξιακή βοήθεια είναι απείρως ε, ανεπαρκή σε σχέση με τις τεράστιες δυσκολίες που έχει η Αφρική. Σε ένα κόσμο ο οποίος έχει βασιστεί, έχει οργανωθεί και διοικείται από το Βορρά. Θα ήταν λοιπόν πιο ενδιαφέρον ένα βιβλίο που να έλεγε. Το πρόβλημα της Αφρικής είναι η επιδοτή στη Γεωργία, για παράδειγμα, ε, στις χώρες του Βορρά στις αναπτυγμένες, ορίστε ένας λόγος για να πούμε ποια είναι τα προβλήματα της Αφρικανικής Γεωργίας, η οποία πήγε στο Βρόντο και σιγά σιγά ε, κατακριμνίστηκε και καταστράφηκε. Και τα παραδείγματα και εξηγήσει είναι άπειρα για να δούμε και να εξηγήσουμε γιατί είναι έτσι ε, η Αφρική και τι πταίει. Δεν λέω ότι δεν φταίνε πολλοί Αφρικανοί, ορισμένοι Αφρικανοί, αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι εκείνος που έχει το λιγότερο φταίξιμο είναι αναπτυξιακή βοήθεια. Και συμφωνώ με τον κύριο Μίτσελ ότι το να γίνονται τέτοιες δηλώσεις δεν βοηθούν. Το μόνο που μπορούν να βοηθήσουν είναι να αποθαρρύνουν, να αποκαρδιώσουν ε, και εκείνους που είναι προσιλωμένοι σε αυτή την προσπάθεια. Εμεί θέλουμε και ε, το κράτος της χώρας μας και ο κόσμος να δίνει περισσότερα στην αναπτυξιακή βοήθεια. Και εδώ βρίσκουν δικαιολογίε για να μην βάζουν το χέρι στην τσέπη και να μειώνεται η βοήθεια και η προσπάθεια αυτή. Αυτό μου φαίνεται ειλικρινά αρνητικό και πολύ λίγο με πίθη ως προς τα επιχειρήματα που βάρα πολύ σύντομα μα παρουσίασε ο συγγραφέας. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Λόβινγκ ότι υπάρχουν και άλλα βιβλία που εκινούν από την αφετηρία ότι προβλήματα υπάρχουν, αλλά δεν καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτό που θα έπρεπε ήταν να γυρίσουμε σε έναν κόσμο αυτοκρατοριών. Δηλαδή αυτός που βοηθάει να ελέγχει κιόλα που πάει βοήθεια και να υπαγρυπνεί και ξέρω εγώ και κυρίω να υπαγορεύει πού θα πρέπει να πάνε τα χρήματα και σε ποιον. Αυτή η σεμνή μου συνεισφορά. Και έχω την αίσθηση ότι έχω χάσει μισή ώρα από τη ζωή μου, κυρία Πρόεδρε. <laughs> Okay. Mais je vais maintenant passer la parole à... Ωραία. Η κυρία Γκάλιντολέν θα πάρει το λόγο. Pour 5 à 7 minutes. Um, yes, thank you. Um... Ευχαριστώ. Ε, στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ανάπτυξη Μένω και ασχολούμαι με το θέμα της αποτελεσματικότητας ε, της ε, βοήθειας. Χάρηκα που άκουσα την παρουσίασή σας, ούτε εγώ το έχω διαβάσει το βιβλίο σας, αλλά βλέποντας τον τίτλο του και ακούγοντας σας σήμερα, Ακούγεται πολύ θετικότερο το μήνυμά σας και ευθυγραμμισμένο με τις δικές μας ε, προσπάθειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Παραδείγματο χάρη, όταν ε, μας μιλάτε για την σημασία των ε, τοπικών ε, κυβερνητικών πολιτικών, ναι, ένα, μία από τις βασικές αρχές είναι η ιδιοκτησία για να είναι αποτελεσματική η βοήθεια και θέλουμε να ενισχύσουμε τη χρήση των ε, κυβερνητικών συστημάτων ε, το ε, μπορεί να προσδιορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση τις πολιτικές της. Τώρα, τι συμβαίνει σήμερα και τι μπορούμε να αλλάξουμε. Άλλο ένα πράγμα που μας απασχολεί ως προς την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Είπατε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Ναι, σε αυτό αποσκοπούμε μέσα από τη διαδικασία κατανομής των εργασιών ε, να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ισότητα στους διάφορους τομείς. Βλέπουμε πώς οι δωρητές δραστηριοποιούνται ε, σε κάθε χώρα για τη διακυβέρνηση, για την εκπαίδευση, ε, αλλά και σε σημαντικότερους τομείς, έτσι, όπως η γεωργία στην οποία αναφερθήκατε και εσείς ε, για να επιτύχουμε λοιπόν έλεγα ισότητα ανάμεσα στις ε, χώρες και να αντιμετωπίσουμε και τις επωνομαζόμενες ορφανές χώρες. Τώρα, να ε, εξηγιάνουμε τις υφιστάμενες δομές. Ναι, και αυτό το επιχειρούμε εναρμονίζοντας τη βοήθειά μας. Δηλαδή, δεν μπορούν όλοι οι δωρητές να κάνουν τα πάντα, ας ειδικευτούμε σε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα και ε, το οποίο θα προσφέρει και μια προσθέμενη αξία στη χώρα που προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Είπατε ότι από πολιτικής πλευράς πρέπει να ε, είμαστε πιο ανοιχτοί, πιο διαφανείς. Ναι, είναι μεγάλη η πρόκληση και μας απασχολεί το θέμα σε όλες τις συζητήσεις που κάνουμε με τα κράτη-μέλη. Ε, αλλά και εδώ λέμε ναι, ας ενσωματώσουμε αυτή την πολιτική διάσταση. Ε, δείτε τι, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατανομή των εργασιών. Ε, ενθαρρύνουμε όλους τους δωρητές να κάνουν μια ανάλυση του συγκριτικού πλεονεκτήματός τους. Αυτή η πολιτική διάσταση ήδη είναι ενταγμένη στο σχέδιο. Φυσικά δεν μπορούμε να την ε, παραμελήσουμε. Θα ήθελα επίσης ε, να σχολιάσετε αν θέλετε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ξέρετε τώρα παρουσιάσαμε το ιαρινό πακέτο με την ε, ανακοίνωση για τους στόχους του χιλιετίας αλλά και ειδικό πακέτο για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας καθώς και για το ρόλο της φορολογίας στην ανάπτυξη. Πολύ θα με ενδιέφερε να σχολιάσετε το έργο μας. Ίσως είχε αλλάξει η εικόνα γιατί το συγγράψατε το 2006 το βιβλίο σας. Μήπως ε, κατά τι έχει αλλάξει η κατάσταση έκτοτε. Ε, βέβαια υπολείπεται. Μεγάλο έργο. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο τώρα στον ε, κύριο Καλντερίση. Σας, θα σας ζητούσα να μην υπερβείτε κατά πολύ το χρόνο που σας αναλογεί πέντε λεπτά δηλαδή συγκεκριμένο. Ευχαριστώ. διάβασα, έγραψα μάλλον το βιβλίο μου, γιατί το, ε, ο στόχος του 0,7% της ε, βοήθειας ε, είναι από τους πιο λανθασμένους στόχους της διεθνής πολιτικής. Για να απαντήσω σε αυτό το θέμα έγραψα το βιβλίο και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, μεγάλος δωρητής αντεξιακής βοήθειας. πρέπει εσείς να γνωρίζετε ότι ο, όγκος της ποιότητας είναι εις της, όγκος της, συγγνώμη, της βοήθειας είναι εις βάρος της ποιότητας της βοήθειας. Ε, για διάφορους λόγους ε, η βοήθεια δεν φτάνει σε αυτούς που την έχουν ανάγκη στους στοχούς. Ε, ε χρειάζεται καλύτερο σχεδιασμός για να φτάσει στους στοχούς. Συμφωνώ ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις μπορεί να δώσουν βοήθεια αποτελεσματική και στο βιβλίο μου μάλιστα πολύ θερμά λέω ότι πρέπει να δίνουμε βοήθεια από τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Τα αποτελέσματα εκεί είναι ξεκάθαρα. Και τα κίνητρα. Ενώ συχνά τα κίνητρα ας πούμε, και τα αποτελέσματα της επίσημης βοήθειας είναι σκοτεινά. Ε, ο τίτλος μου δεν είναι ε, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει η βοήθεια στην Αφρική είναι ότι δεν λειτουργεί απλώς. Ε, εγώ, ας πούμε, ε, διαπίστωσα ότι στην, σε άλλες περιοχές του, του κόσμου, όπως στην Ινδονησία, ας πούμε, που ήμουν επί 8 χρόνια, μια χαρά τα πάει η βοήθεια. Είναι πολύ αποτελεσματική και βοηθάει τους αγρότες για να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Ε, επίσης στο βιβλίο ε, λέω και θετικά πράγματα ε, για το Μαυρίκιο, την Ποτσουάνα, η Γκάνα, η Μοζαμβίκη, η Ουγκάντα, η Τανζανία. Βέβαια με κάποιες παλινοδίες, με κάποιες δυσκολίες μέσα σε 15-20 χρόνια τελικά πήραν σωστές οικονομικές αποφάσεις και βελτίωσαν τους πόρους τους. Χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικό τρόπο τους πόρους τους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι καθόλου βοήθεια είναι καλύτερα από ένα μια άφθονη ας πούμε βοήθεια. Εγώ απλώς λέω ότι θα πρέπει να διδαχθούμε ε, από τα μαθήματα των τελευταίων 45 ετών και να ανακατευθύνουμε σε νέα προγράμματα τη βοήθεια. Αυτό που είπατε ε, για μια άλλη συγγραφέα είναι απλουστευτικό. Ε, ότι υπάρχει μια επιλογή ανάμεσα στην, στις ξένες επενδύσεις ας πούμε και στην ξένη βοήθεια ή το ένα ή το άλλο. Κανένας δεν πιστεύει ότι η ξένη βοήθεια θα δημιουργήσει ανάπτυξη. Ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί, εφαρμόζεται μάλλον σε τομείς όπου δεν υπάρχει τοπική γνώση, δεν υπάρχει παρέμβαση της κυβέρνησης κτλ. απλώς θα πρέπει να εστιάσει καλύτερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επίση, το εμπόριο φυσικά είναι πολύ πιο σημαντικό από τη βοήθεια για να βοηθήσει τον κόσμο να βγει από τη φτώχεια. Αυτό είναι γεγονό, είναι αναφυσβήτητο. Ανέφερα και τη γεωργία στην αρχική μου παρέμβαση επίτηδε, γιατί στην Αφρική παραμένει ε, ο βασικός τομέα πλούτου. Κι όμως οι κυβερνήσεις ε, την ξεχνάνε. Ξεχνούν, α πούμε, ότι οι δικέ μα κυβερνήσει, α πούμε στον Καναδά, στι ΗΠΑ, στη Βραζιλία κτλ. κέρδισαν πάρα πολλά από τη Γεωργία. Στην Αφρική την παραμελούν. Ε, Μία χώρα σαν το Τσάντ δεν μπορεί να βοηθηθεί από την βοήθεια, όπου οι γεωργοί δεν δίνουν, ας πούμε, δεν βάζουν λιπάσματα στι βασικέ οδιέ του. αν μένουν 100 μέτρα από το δρόμο. Ε, γιατί α, αν είναι πολύ κοντά στο δρόμο, τα, φορτηγά του στρατού σταματάνε το, τη νύχτα και κλέβουν τους καρπούς, κλέβουν ας πούμε τις τα λοιπά Οι δυνάμεις ασφαλείας. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα, πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Ε, συμφωνώ. Ότι όταν είπα για τους επιθεωρητές, ας πούμε, ε, δεν λέω κάτι καινούριο. Από τις διάφορες ε, μεθόδους που χρησιμοποίησαμε στο παρελθόν, ακόμη και αποστολές ας πούμε εποπτείας της Παγκόσμιας Τράπεζας που όλοι θεωρούμε ότι είναι σωστές, ε, κάθε 6 μήνες τις θέλουμε για 2-3 μέρες ας πούμε αυτές οι αποστολές. Δεν αρκούν αυτά τα πράγματα. Είναι αραιή αυτή η επιθεώρηση. Εγώ θέλω να γίνεται πιο συχνά, πιο μόνιμα από τους Αφρικανούς, οι δυνατόν. Ε, και θα μπορούσαν Αφρικανοί να επιστρέψουν στις χώρες τους για να κάνουν μια τέτοια, ένα τέτοιο ευγενές ας πούμε, έργο που θα έχει και καλύτερες, καλύτερους όρους ας πούμε, απασχόλησης. Επίσης δεν λέω να μην βοηθήσουμε ας πούμε, με συμπληρώμα εισοδήματο φτωχού. Επίσης, εγώ γνωρίζω το πώς λειτουργεί το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ξεκίνησα την καριέρα μου. Ε, Πιστεύω ότι ο, αν κάποιος έχει αποδείξει ότι λειτουργεί αποτελεσματικά, θα πρέπει να, να ανταμείβεται. Παραδείγματο χάρη να δούμε, ας πούμε, χώρες όπως το Τσάντ και άλλες χώρες της Αφρικής, τι ποσοστό παιδιών πηγαίνουν στο σχολείο ή κοριτσιών κτλ. Ε, πόσο υλοποιούνται οι στόχοι και μετά από δύο-τρία χρόνια ε, κάνουμε μια αποτίμηση. Για άλλες χώρες όμως χρειάζονται ας πούμε ε, εποπτεία κατά τη διάρκεια των εκλογών. Διεθνή εποπτεία κατά τη διάρκεια των εκλογών και θα πρέπει να το δεχθούν αυτό, θα πρέπει να δεχθούν τέτοιους όρους. Ε, πρέπει να δούμε, εν από χώρα σε χώρα και να προσαρμοστούμε ανάλογα με την κατάσταση εκάστοτε χώρα. Ευχαριστώ. Θα πάμε στο σημείο 9. Έχουμε τώρα την παρουσίαση του προγράμματος δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για ε, την υλοποίηση των κανονισμών για τα δάση, τη διαχείριση και τις εμπορικές συναλλαγές FLEGT για την παράνομη υλοτομία και ε, το εμπόριο που απορρέει αυτή και πώς θα καταπολεμηθεί για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη δυνατότητα των κρατών ε, που παράγουν ε, ξυλία να διαχειριστούν την ξυλία αυτή. Έχουμε τον κύριο Ριέρα ενώπιόν μας που είναι διευθυντής ε, στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μας παρουσιάσει τις εθελοντικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες. Έχετε το λόγο για ένα τέταρτο της ώρας, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Σριέρα. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε εδώ ε, πώς έχει το πρόγραμμα δράσης FLECT ε, αυτό τον καιρό και να σας ε, δείσουμε ε, ακριβώς ε, τη σημασία του προγράμματος, το οποία γνωρίζετε και εσείς ε, ως νεοσύστατη ε, Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, θα χρειαστούμε και καλωσορίζουμε τη διαρκή σας υποστήριξη. Γιατί παρουσιάζουμε σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα δράσης FLECT και πού βρισκόμαστε σήμερα. Να σας πω, διότι έχουμε ήδη τρεις ε, συμφωνίες εταιρική σχέσης ε, που έχουν ολοκληρωθεί ε, και η μία έχει υπογραφεί και έχει κυρωθεί κιόλας στην περίπτωση της Γκάνας. Το Κονγκό είναι στη διαδικασία κύρωσης και το Καμερούν τον άλλο μήνα μονογράφεται η συμφωνία. Και διαπραγματευόμαστε πολλά προγράμματα αυτό τον καιρό και με τη Λιβύρια και τη Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής και σύντομα θα αρχίσουν οι πραγματεύσεις με την Καμπόν και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και επίσης και με την Ινδονησία και τη Μαλαισία διαπραγματευόμαστε. Και δεχόμαστε και αιτήσει εκδήλωση ενδιαφέροντος και από τη Λατινική Αμερική. Βεβαίως, ε, ε, η εισαγωγή ξυλία από τη Λατινική Αμερική στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μικρότερη. Ε, ωστόσο, η αγορά της Λατινικής Αμερικής ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για τη διαδικασία αυτή και έχουν διεξαχθεί και πολλές αποστολές στην Λατινική Αμερική για να ενημερωθούμε. Είναι μια πολύ απλή ιδέα αυτή οι χώρες που παράγουν ξυλία εξάγουν ξυλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα σύστημα πιστοποίησης ε, που διαβεβαιώνει τους Ευρωπαίους καταναλωτές ότι η ξυλία αυτή είναι νόμιμη και δεν είναι προϊόν λαθρέας υλοτόμησης και κυκλοφορεί κανονικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν μια κατάσταση που είναι προς και των δύο μερών και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ε, ε, είναι ήσυχοι ότι η ξυλία αυτή είναι νόμιμη και ο τρόπος με τον οποίο ε, συλλέγεται και ο τρόπος με τον οποίο εξάγεται και αυτό είναι θετικό για τις αναπτυσσόμενες χώρες και την ανάπτυξη της κάθε χώρας το να καθησυχάζουμε τον καταναλωτή και βεβαίως και είναι προς όφελος και της ίδιας της χώρας ότι θα έχει πρόσβαση στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι μπορούμε καλύτερα να διαχειρίζονται τα δάση τους. Ε, είναι απλή η αρχή που κρύβεται από πίσω ε, στη θεωρία, αλλά όταν φτάνουμε στις διαπραγματεύσεις καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι πολύ πιο περίπλοκη η κατάσταση. Η παρανομία δεν οφείλεται πάντα στους ίδιους λόγους σε όλες τις χώρες. Μπορεί να παρανομούν για πολύ διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή η δυνατότητα, η αδυναμία του κράτους, ε, φορολόγησης, ε, άλλα θέματα διαχείρισης των δασών και επίσης όπως ε, μάλλον η κατεύθυνση εισαγωγών-εξαγωγών είναι απλή. Ε, Όπω θα μπορούσε κανεί να φανταστεί, δεν έχουμε άμεσε εξαγωγέ. Α πούμε, έχει κάποιο ξυλία και την εξάγει προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και φτάνει στον τελικό καταναλωτή. Είναι ολόκληρη αλυσίδα η εξαγωγή τη ξυλία και το εμπόριο σε όλο τον κόσμο. Όπως άλλωστε συμβαίνει και με οποιοδήποτε άλλο αγαθό και έχουμε εισαγωγές και εξαγωγές από διάφορες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έμεσα. Εξάγεται σε μια άλλη χώρα πρώτα το ξύλο και μετά φτάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαχείριση των δασών τώρα. Η δασοπονία είναι μια ιστορία ε, περίπλοκη. Σκεφτείτε και μόνο πόσοι ενέχονται στη διαχείριση των δασών με πολύ ειδικά συμφέροντα και πολύ αποκλίνοντα συμφέροντα. Δεν είναι μόνο τα συμφέροντα των παραγωγών, των καταναλωτών και οι κυβερνήσεις και οι διάφορες ε, ε, εταιρείε μεσάζοντες ή εκείνοι που ε, ζουν στην Ήπεθρο εκείνοι που επεξεργάζονται το ξύλο και εξάγουν ε, ή εκείνοι που παράγουν για την εντόπια αγορά της κάθε χώρας ή για τις εξαγωγές, για την παγκόσμια αγορά. Είναι λοιπόν μια κατάσταση περίπλοκη, ένας περίπλοκος κλάδος έτσι κι αλλιώς ε, της οικονομίας και ζωτική σημασίας από πλευράς εισοδήματος για πολλές χώρες. Οπότε μπαίνουν και άλλα περίπλοκα ζητήματα που δεν είναι εύκολο να ε, συμφιλειωθούν. Η πρώτη συμφωνία που έχει κυρωθεί ήδη με την Κάνα μας δίδαξε πολλά σημαντικά και ε, πολύτιμα για τις διαπραγματεύσεις που κάνουμε αυτόν τον καιρό με άλλες χώρες. Αλλά βεβαίως η πραγματικότητα διαφέρει από χώρα σε χώρα και από πλευρά θεσμών και από πλευρά εμπορίου. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μία συμφωνία που να συνάπτουμε την ίδια ακριβώ με όλε τι χώρε. Η ε, συμφωνία λοιπόν που επιτεύχθηκε με την Κάνα είναι ένα πλαίσιο χρήσιμο και ε, πηξίδα για τις επόμενες διαπραγματεύσεις με τη Λιβυρία ας πούμε αρχίσαμε πριν από ένα μήνα και το γεγονός ότι ε, έχουμε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι χρήσιμο και μας βοηθάει για τις επόμενες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Τώρα, ποια είναι αυτά τα διδάγματα. Ε, ε, θα τα ξεχώριζα στα διαδικαστικά και στα ουσιαστικά. Ε, ως προς τον τύπο τώρα και τη διαδικασία. Οι συμφωνίες αυτές FLECT μας επέτρεψαν να συζητούμε θέματα διαχείρισης δασών με ένα ευρύτερο φάσμα ε, ενδιαφερομένων στην ίδια τη χώρα και την κυβέρνηση της χώρας. Στο παρελθόν συζητούσαμε για τα δάση με ε, τα Υπουργεία Δασών. Το γεγονός όμως ότι αυτή η συμφωνία κυρίως εμπορική οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικέ σχέσης. Ε, συζητάμε και με Υπουργείο Εμπορίου, Υπουργείο Αναπτύξη Πέθρου, Υπουργείο Οικονομικών ε, και όχι μόνο με τη δασική υπηρεσία σε κυβερνητικό επίπεδο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, συζητούμε με πολλούς ενδιαφερομένους και από τις κυβερνήσεις και από τις χώρες αυτές. Στη συνέχεια, ε, μας απασχολούν θέματα που άπτονται της κυριαρχίας των κρατών, έτσι. Και έχουν ε, μεγάλη πολιτική ευαισθησία. Όταν συζητάς αν προσφέρεται έναν καλό ένα νόμο ή αν είναι αρκετά αυστηροί οι μηχανισμοί κυρώσεων και προστήμων για εκείνου που δεν συμμορφώνονται. Όταν μπαίνουμε σε τέτοια ζητήματα, θίγονται άμεσα ε, θέματα κυριαρχίας των κρατών. Ε, στη συνέχεια, όχι μόνο διευρύναμε τις συζητήσει που έχουμε στο εσωτερικό των κυβερνήσεων, αλλά συμμετέχουν και άλλοι, ε, όπως είπαμε, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΙΟΜ, και εκπρόσωποι ε, του κλάδου ε, της ξυλίας. Είναι πολύ χρήσιμη ε, πραγματικά αυτή η διαδικασία, σας διαβεβαιώ. Αυτό το είδαμε όταν επισκεφτήκαμε τις διάφορες χώρες. Είχαμε τις διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με πάρα πολλές χώρες με κλάδους ενδιαφερμένων πολλού. Και οι κυβερνήσεις πλέον έχουν καταλάβει ότι αξίζει τον κόπο να γίνονται αυτές οι ζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις. Βεβαίως λίγο επιβραδύνεται η διαπραγμάτευση με όλη αυτή τη διαβούλευση, αλλά τελικά μας βοηθάει γιατί οι τελικές συμφωνίες είναι πολύ πιο ουσιαστικές και πιο ε, ισχυρές. Έρχομαι τώρα στην ουσία. Ποια είναι τα διδάγματα. Βοηθήσαμε και τις χώρες τις ίδιες να ξεκαθαρίσουν το νομοθετικό τους πλαίσιο και τις βοηθούμε να ε, κάνουν μια αξιολόγηση οι ίδιες για το πόσο ε, ισχυρό είναι το νομοθετικό τους πλαίσιο, πόσο καλή είναι η νομοθεσία τους, τους βοηθάμε Επίσης, νομίζω ε, να έχουν και τις νομικές εγγύησεις που χρειάζονται για να μειώνεται η διαφθορά και να βελτιώνεται η επιβολή του νόμου. Όλες αυτές οι συζητήσεις επίσης γίνονται και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με τον ιδιωτικό τομέα εκτός από τις κυβερνήσεις και αυτό μας βοήθησε επίσης πάρα πολύ. Και τέλος πιστεύω ότι βοηθήσαμε τις χώρες να κάνουν μεγάλες πρόοδους στη διαφάνεια ε, και στην πρόσβαση στην ενημέρωση, διότι ακριβώς συμμετείχαν πολλοί εταίροι στη διαπραγμάτευση. Τέλος, για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι ίδιες οι χώρες ακριβώς μετά από πίεση ε, ε, τις βιομηχανίες στο εσωτερικό, όπως στο Κονγκό και στη Γκάνα και στο Καμερούν, ε, ζήτησαν οι συμφωνίες να μην διέπουν μόνο τις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και προς άλλες αγορές. Και όχι μόνο για τις εξαγωγές, αλλά και για την παραγωγή που προορίζεται στην αχώρια κατανάλωση. Ισχύει αυτό. Οι διάφοροι λοιπόν ενδιαφερόμενοι Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ε, πρόβαλαν τις θέσεις τους ακριβώς για να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία που να ισχύει προς όλους. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής. Άριστη συνεργασία είχαμε με τα κράτη-μέλη, τα οποία απουσιάζουν μάλλον σήμερα. Γι' αυτό χαίρομαι ακόμα περισσότερο που μπορώ να το πω και εν τη απουσία τους είχαμε υποστήριξη από διάφορες χώρες σε διαφορετικές διαδικασίες. Ας πούμε, στην Κάνα μας βοήθησε το Ηνωμένο Βασίλειο και οι 100 χώρες. Ε, σε άλλες περιπτώσεις η Γερμανία, η Γαλλία, οι άλλοι. Χωρίς αυτή την υποστήριξη, αυτή την όθηση από τα κράτη-μέλη, Ε, θα χρειαζόταν ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιτύχουμε τις συμφωνίες αυτές. Λοιπόν, η διαδικασία αυτή αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί. Νομίζω τώρα αποκτά κάποια ορμή και φόρα. Η καλή διακυβέρνηση και η διαφανής διακυβέρνηση σε ένα τόσο κρίσιμο και περίπλοκο τομέα όπως είναι η ε, υλοτόμηση των δασών είναι μια καλή αρχή, έτσι ώστε να υπάρχει καλή διακυβέρνηση και ε, διαχείριση σε όλους τους άλλους τομείς. Και έχουμε ακριβώς και θετική επίδραση των συμφωνιών αυτών και προς άλλους κλάδους. Και δείχνει αυτό ότι εφόσον εφαρμόζεται εδώ και είναι καλό, μπορεί να επεκταθεί και αλλού. Είναι καλή λοιπόν αρχή και ένα καλό παράδειγμα και για άλλους κλάδους της οικονομίας. Ένα τελευταίο Η διαδικασία αυτή απαιτεί ε, κάποιες προσπάθειες βεβαίως και από πλευρά των κρατών αυτών έτσι, για να μπορέσουν να είναι στο επίπεδο των προτύπων και προδιαγραφών που απαιτούνται. Χρειάζεται μια ολόκληρη αλυσίδα να στηθεί παρακολούθηση, συνοδείας, ελέγχου από την αρχή, από το δέντρο μέχρι ε, το τελικό προϊόν. Ε, είναι μια διαδικασία περίπλοκη και χρειάζεται και κάποια τεχνική υποστήριξη και από εμά και από άλλους δωρητές. Και προσβλέπουμε εν ευθέτω χρόνο να μας υποστηρίξετε κι εσείς αν χρειαστεί ε, επιπλέον ενίσχυση προς τις χώρες αυτές για να ανταποκριθούν στο έργο τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρτίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Και ευχαριστώ τον κύριο Ριέρα για τις πληροφορίε που μας έδωσε για το θέμα αυτό. Πρέπει να συγχαρούμε την Κομισιόν. Ε, πρέπει να γίνει πιο γνωστή αυτή η πρωτοβουλία. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πολύ λίγοι συναδελφοί είναι ενημερωμένοι για αυτά τα προγράμματα, για αυτές τις ε, πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και ένα σχόλιο. Η ερώτηση είναι η εξής. Πώς θα κινητοποιηθούμε, ε, πώς θα κινητοποιήσουμε κάποιες χώρες για να προσυπογράψουν αυτούς τους στόχους. Τι συμφέρον έχουν αυτές οι χώρες να συμμετάσχουν. Παραδείγματο χάρη, οι εταιρείε που κόφουν το ξύλο και το βάζουν στο εμπόριο, α πούμε, ε, κερδίζουν πάρα πολλά. Τι μπορούμε να προσφέρουμε εμεί ε, στι κυβερνήσεις για να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία, ε, μια συμφωνία μαζί μας. Δηλαδή να του προσφέρουμε εμεί κάτι παραπάνω από αυτά που του δίνουν οι εταιρείε. Πώ μπορούμε να τι κινητοποιήσουμε. Τώρα ένα σχόλιο. Να σα μιλήσω για μια εμπειρία μου. Μια εμπειρία μου. Με ελικόπτερο πήγα από τα σύνορα της Βενεζουέλας προς το εσωτερικό της Βραζιλίας. Δηλαδή Ουσιαστικά είναι ε, τα δάση του Αμαζονίου εκεί, που διάφορες χώρες ε, συνεργάζονται. Στη Βενεζουέλα η κυβερνητική πολιτική διατηρεί ε, το δάσος του Αμαζονίου σχεδόν παρθένο. Περνάει κανείς τα σύνορα και άμα το δει κανεί από πέρσι μέχρι φέτο, χιλιόμετρο χιλιόμετρο φαίνεται, ή ξέρω εγώ, εκατοντάδε χιλιόμετρα επί εκατοντάδε, μπαίνοντα στη Βραζιλία, κόβουν. Και ε, με τρόπο πραγματικά πάρα πολύ βίαιο, εκτάρια ολόκληρα. Με ελικόπτερο το βλέπει κανείς καλύτερα γιατί περίπταται και το βλέπει από κάτω και περνάει από το δάσος σε μια πράσινη σαβάνα, έτσι, ένα τέτοιο είδος, όπου κάποτε ήταν δάσος και αν ξαναπετάξεις μετά από δύο μήνες έχει πάει 50 χιλιόμετρα πιο πέρα η αποψήλωση. Και σας μιλάω τώρα για ε, ένα πλάτος 40 χιλιόμετρων, έτσι, το οποίο βαθαίνει μήνα με το μήνα και κόβει το δάσος του Αμαζονίου. Και θα εξαφανιστεί το παρθένο δάσος εκεί. Λοιπόν, απέναντι σε τέτοιες δράσεις μεγάλων κρατών τι κάνεις. Εγώ το συζήτησα με τις βραζιλιανικές αρχές όπως και πολλοί συνάδελφοι, είναι και δικοί μου φίλοι. Μου λένε ότι ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε οι εταιρείε και τα λοιπά, ξυλίας, ε, είναι ανεξέλεγκτες στη δράση τους. Ή ε, έχουν τέτοια κέρδη που και είναι και τόσο υποφελές διότι ε, επιτρέπουν την εκτατική κτηνοτροφία γιατί ανοίγουν μεγάλες εκτάσεις και ρωτάω, εσεί τι κάνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταλάβουν οι χώρε ότι δεν είναι μόνο ε, ε αυτό το όφελος ότι δεν χαλάνε το δασο, αλλά έχουν και συγκεκριμένα ωφέλη από μια λελογισμένη εκμετάλλευση των δασών χωρίς να τα εξολοθρεύουν και να τα καταστρέφουν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και κύριε Ρία. Ευχαριστούμε ο κύριο Μίτσελ. Ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τον συνάδελφο Μαρτίνες. Και ευχαριστώ την Επιτροπή για την παρουσίαση. Είναι πολυσχηδή τα ζητήματα, τα αναπτυξιακά. Δύσκολα μπορεί κάποιος να τα παρακολουθεί όλα και να παραμένει ενήμερος. Ε, και έχουμε και πάρα πολλές ε, ε, ανησυχίες ούτως ή άλλως για τα ζητήματα που σχετίζονται με το κλίμα. Λοιπόν, η Γκάνα τι κερδίζει από μια τέτοια συμφωνία και οι υπόλοιπε χώρες, δηλαδή πώς ακριβώς τους πουλάτε τις συμφωνίες, τι τους υπόσχεστε. Στο παράρτημα για την Γκάνα λέει ότι δίνει αναπτυξιακή βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη ενδογενών ικανοτήτων για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Στην περίπτωση της Γκάνας ε, αυτό γίνεται μέσα από έναν ε, ε, μηχανισμό του δημοσιονομικού πολλαπλών δωρητών. Άντε να το εξηγήσει αυτό σε κάποιον που σε ψηφίζει. Τέλος πάντων. Ε, τι ακριβώς σημαίνει αυτό, ποιο, πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, ε, και για την ανάπτυξη ενδογενών Τέλο πάνω καλή τύχη, γιατί φαίνεται να είναι ενδιαφέρον αυτό που κάνετε. Ε, ευχαριστούμε. Κάτι άλλο, υπάρχει άλλη ερώτηση. Όχι. Παρακαλώ. Thank you, thank you, I mean... Ευχαριστώ. και τον κύριο Μαρτίνε και τον κύριο Μίτσελ ε, για τα καλά τους λόγια και για τις ερωτήσεις τους. Η πρώτη ερώτηση του κυρίου Μαρτίνες ε, και η ερώτηση του κυρίου Μίτσελ νομίζω παρουσιάζουν κοινά σημεία. Τι συμφέρον έχουν ε, οι εν λόγω χώρες, ήταν το ερώτημα. Σίγουρα η ευρωπαϊκή αγορά και όχι μόνο έτσι για τα προϊόντα δασοκομείας ε, ε, γνωρίζει σημαντικές αλλαγές. Και με τις δράσεις αυτές αυξάνεται η ανησυχία που νιώθουν οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αν είναι νόμιμο το ξύλο που αγοράζουν άμεσα, κυρίως έμεσα από αυτές τις ε, χώρες και από δάση που αποψηλώνονται. Λοιπόν, μακροπρόθεσμα, όσε χώρε έχουν υπογράψει τέτοιες ε, συμφωνίε εθελοντική εταιρική σχέση. θα έχουν πλεονέκτημα στην αγορά. Τι εννοώ, θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε αυτές τις αγορές υποθετικά βέβαια. Γιατί θα έχετε δει δημοσιεύματα στον τύπο σχετικά με τι αλλαγέ που σα είπα πώ σημειώνονται στι αγορέ. Το 2011 ελπίζουμε να μπορέσουμε να εισάγουμε το πρώτο ξύλο πιστοποιημένο φλέκτ ε, από αυτές τις χώρες. Και τότε θα είναι η σωστή στιγμή να γίνει εκστρατεία ενημερωτική με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την όλη διαδικασία. Για να δοθούν ε, ε, κάποια ειχέγγυα σε όλους μας για τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Αυτό ήταν ένα πρώτο στοιχείο. Δεύτερον, τι κερδίζει η Γκάνα, με ρωτήσατε. Αν μπορούμε να μειώσουμε τα έσοδα από την παράνομη λοτομία και να αυξήσουμε την ικανότητα της κάθε χώρας να αναπτύξει ε, το τομέα αυτό ναι, είναι καλό. Η Λιβυρία παραδείγματο χάρη πριν τον εμφύλιο πόλεμο και τις ε, αναταραχές ε, ήταν βασικός τομέας η δασοκομεία τώρα, είναι μηδενικά τα έσοδα. Δηλαδή τους βοηθούμε για να βάλουν τάξη στον κλάδο αυτό και να έχουν καλύτερη διακυβέρνηση. Για να έχει καλύτερο δυναμικό αυτός ο κλάδος, καλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό δηλαδή. Βραζιλία, Βενεζουέλα, Νομίζω ότι αυτό μπορεί να μας δείξει τι μπορεί να συμβεί σε άλλες χώρες όπως στην Κάνα ή στην ακτή του Ελεφαντοστού. Αν η Γκάνα εισέλθει σε αυτή τη διαδικασία της καλύτερης ε, διακυβέρνησης, ελοχεύει λοιπόν αυτός ο κίνδυνος να περνάει το ξύλο από την ακτή του Ελεφαντοστού μέσα από την Γκάνα. Αυτό προβλέπεται όμως στη συμφωνία. Υπάρχει σχετική ρήτρα για να το αποφύγουμε. να λάβαμε αυτή την πρωτοβουλία για να ε, αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο. Γι' αυτό μιλάμε για τη δέουσα ε, νομική παρακολούθηση ε, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, σε εισαγωγές θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση ότι δεν έχει υλοτομηθεί παρανόμως η ξυλία. Σε αυτή την πρόταση λοιπόν ε, ε, για την ε, δέουσα επιμέλεια, due diligence, θα την αναλύσετε εξάλλου σύντομα. Θα δείτε ότι σε κάθε συμφωνία FLECT πληρείται αυτό το κριτήριο, αυτή η ρήτρα για τη δέουσα επιμέλεια. στις αφρικανικές χώρες βέβαια δεν βλέπουν ε, ε, με τον ίδιο τρόπο αυτό το πρόβλημα. Δεν αντιλαμβάνουν την τραγωδία με τον ίδιο τρόπο. Κύριε Μίτσελ, αυτός ο δημοσιονομικός ε, μηχανισμός πολλαπλών δωρητών υπάρχει στο περιβαλλοντικό τομέα, στην Κάνα και τι θα υποστηρίξουμε μέσα από αυτό το μηχανισμό. Αυτό θα είναι συνάρτηση ε, των αναγκών κάθε χώρας. Ε, ο Υπουργός Περιβάλλοντος προσπαθεί να πείσει τον Υπουργό Οικονομικών ε, στην Κάνα ότι αξίζει αυτή η συμφωνία. Ότι δηλαδή μέσα από αυτό τον δημοσιονομικό μηχανισμό ανατομέα θα έχουμε αυτήν την αλυσίδα επιμέλειας, αλυσίδα ελέγχου είναι σημαντικό αυτό γιατί χρειάζεται και η χνηλασιμότητα. Το ξύλο περνάει από πάρα πολλά στάδια μέχρι να εξαχθεί. Οπότε στην Κάνα πέρα από την ενίσχυση της ε, τεχνικής ε, ικανότητας της Δασοκομικής Επιτροπής ε, θα συγκροτήσουμε αυτόν τον μηχανισμό παρακολούθησης και θα υποστηρίξουμε τη λήψη αποφάσεων σε κυβερνητικό επίπεδο. Γιατί υπάρχει ειδική συμφωνία για αυτό το θέμα. Στο θεματικό πρόγραμμα περιβάλλον παρέχουμε τεχνική αρρωγή ενισχύοντας ε, ε, τις, ε, τα, τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες ε, γιατί αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκη αυτή η διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω ε, για την συνεργασία. Μπορείτε να